Οπότε μέχρι να έρθει πρέπει να έχουμε λύσει τα προβλήματα. Επειδή είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων, έστω και καθυστερημένα, εύχομαι στους παρόντες, διερμηνείς, υπαλλήλου και φυσικά τους συναδέλφους βουλευτές τις καλύτερες μου ευχές. Παρακαλώ την πτέρυγα των πολιτικών ομάδων να σοπάσει. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης και προτείνω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με τις εξής ελεγές. Πρώτο, Πού είναι αλήθεια έκθεση της κυρίας Γκρελιέ που είχαμε για σήμερα το πρωί Ο κύριος Γκάλαχερ ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος και δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα το πρωί, οπότε το αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση. Πρέπει όμως να μιλήσω και με την κυρία Γκρελιέ για το τελικό χρονοδιάγραμμα. Πάντως αύριο δεν θα εξετάσουμε την έκθεση της κυρίας Γκρελιέ. Μα πού την έχω αλήθεια εγώ την ημερήσια διάταξη σήμερα και δεν την βρίσκω. στο τελευταίο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης που είναι για τα οικονομικά για τον προπολογισμό. Α, μάλιστα. Το τελευταίο σημείο για την ολοκληρωμένη αλληλεία, η κυρία Πατράο είναι άρρωστη. Οπότε θα πάει το σημείο 13 στη θέση του 8 που είναι η έκθεση σχετικά με την ετήσια συνεδρία της Επιτροπής Αλίας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού στη Χονολουλού. Λοιπόν, πρακτικά της 30ης Νοεμβρίου και της 1ης Δεκεμβρίου τα οποία θα εγκριθούν ανακοινώσεις του, της Προέδρου δεν έχω τίποτα να σας πω και πάμε στο τέταρτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι οι ανταλλαγές απόψεων με τον κύριο Φαζέκας ο οποίος είναι ο Ούγγρος υπουργό για την ανάπτυξη της Υπέθρου και είναι ο Προεδρεύων, τον οποίο βλέπω να καταφθάνει. Να το χαιρετήσω λοιπόν.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 Okay. Bueno, eh, en primer lugar, eh, eh, damos eh, Καλώς ορίζουμε τον κύριο Σάντορ Φαζέκα, είναι Ούγγρος Υπουργός Ανάπτυξης ε, της Υπέθρου και Προεδρεύων του Συμβουλίου και θα μας μιλήσει για τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας. Καταρχήν κύριε Πρόεδρε να σας ε, καλωσορίσω και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για το εξάμεινο της Ουγγρικής Προεδρίας. Ευελπιστούμε να ε, ε, μπορέσετε να πεγκλωβίσετε πολλά θέματα που εκκρεμούν στην Επιτροπή Ελίας. Εγώ πριν σας δώσω το λόγο και φυσικά μετά θα έχουμε κοινή συζήτηση με όλους τους βουλευτές θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία τα οποία θεωρώ ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε αυτή την Επιτροπή. Πρώτο, είναι η μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Όπως ξέρετε έπρεπε καταρχήν να παρουσιαστούν οι προτάσεις της Κομισιόν. Δεν έχει όμως οριστεί ε, τελειωτικά το χρονοδιάγραμμα και ελπίζουμε ότι εσείς θα μπορέσετε να ασκήσετε πιέσεις στην Κομισιόν ούτως ώστε οι προτάσεις αυτές να εμφανιστούν στο τραπέζι υπό την Προεδρία σας και να τις συζητήσουμε. Μετά υπάρχει ένα θέμα που ανησυχεί ιδιαίτερα αυτήν την Επιτροπή και είναι τα σχέδια διαχείρισης όπως ε, ξέρετε εμείς ε, έχουμε μπλοκάρει δύο σχέδια, είναι για την, ε, για την Ατσούγα και και περιμένουμε να βρεθεί μία λύση όπως ε, επίσης ε, και το σχέδιο για τον μπακαλιάρο, το μερλούκιο του Βορρά που ελπίζουμε να βρεθεί μία λύση με ε, μία, λύση που θα μας ικανοποιήσει όλους. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι η συμφωνία, η ελευτική συμφωνία με το Μαρόκο που θα λήξει στις 27 Φεβρουαρίου και κανένας δεν λέει τίποτα προς στιγμήν. Υπάρχουν τώρα εδώ διαφορετικές θέσεις. Είναι αυτοί που θέλουν να συναπαρατείνουν τη συμφωνία, άλλοι που δεν θέλουν. Ε, αλλά δεν έχει δοθεί καμία προπτική. Και έχουμε εμείς ε, όλοι ε, όλο τον αλλιευτικό μας στόλο ε, που θα πρέπει να βγει από αυτήν τη ζώνη και δεν έχουμε ιδέα ακόμα για τίποτα. Η Κομισιόν είναι πολύ πιο ευέλικτη από μας. Και να σας πω το εξής. Εγώ συμμετείχα ως παρατηρήτρια στην Επιτροπή Αιδείας Δυτικού και Κεντρικού Ηρωνιειδηνικού στη Χονολουλού. Πήγα στη Χονολουλού, πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη στη Χονολουλού. Έκανα τη δουλειά μου ως εκπρόσωπος και μου έρχεται όμως μετά τις διακοπές μία επιστολή που λένε ότι δεν επιτρέπουν στην κυρία Φράγκα να συμμετέχει ως παρατηρήτρια στην συνεδρίαση στη Χονολουλού. Βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργούν τα πράγματα σήμερα. Εμείς ελπίζουμε πολλά σε εσά δεν... Δεν χρειάζεται κανείς να είναι υπουργό μιας μεγάλης αλληλευτικής χώρας για να είναι ένας καλός υπουργό αλλίας. Ελπίζουμε λοιπόν πολλά σε εσά, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα μας πείτε και οι συνάδελφοι θα σας θέσουν τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ε, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας και καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για τα εισαγωγικά σχόλια. Ε, τα θέματα της αλίας και η σημασία της αλίας κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετική σημασίας και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα παρακολουθήσω από κοντά αυτές τις πολιτικές κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Η Ουγγρική Προεδρία βλέπει αυτά τα θέματα όχι μόνο από τη σκοπιά της οικονομίας. Η αλληλεία και η υδατοκαλλιέργεια αφορά τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη. Εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και διαβίωση Η πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα μου δεν έχει πολύ μακρά παράδοση σε θέματα ε, αλίας και θαλάσσιας πολιτικής. Αυτό είναι αληθές. Ωστόσο, τούτο μπορεί να είναι πλεονέκτημα ε, διότι βλέπει κανείς τα πράγματα έξωθεν όταν δεν επηρεάζεται άμεσα από τα γεγονότα. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής αλίας είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας. Μία από τις ε, βασικές μας προτεραιότητες είναι η βιωσιμότητα, η αηφορία της πολιτικής. Αυτή είναι μία από τις προτεραιότητες μας. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι η Ουγγρική Προεδρία θα διώξει να συνεργαστεί με, την, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ στενά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, δουλεύουμε μαζί με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας και χαίρομαι για τη συνεργασία με σας. Ε, ελπίζω ότι μαζί θα μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα στην ε, επεξεργασία της νομοθεσίας. Για την ε, διαβούλευση τώρα. Μιλάω για την διαβούλευση. Πριν μιλήσω για το πρόγραμμα της Προεδρίας, να ευχαριστήσω τον Κρίς ε, Πέτερς που ήταν ο προκάτοχός μου για την εξαιρετή εργασία, εργασία του. Υπάρχει παρεμβολή από κινητά τηλέφωνα και δεν ακούν οι διερμηνείς. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας ε, ήταν τρεις βασικοί, τα βασικά θέματα που εξετάστηκαν και επιτεύχθηκαν στην νομοθετική διαδικασία. Έχουμε κάποια θέματα λοιπόν ε, για την αλληλεία στο Συμβούλιο του Απριλίου και, της, και του Ιουνίου. Είναι ε, η αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής ε, πολιτικής. Το πολιετές, τα πολιετή σχέδια διαχείρισης και η συνέχιση της συνθήκης της Λισαβόνας με μια σειρά θεμάτων. Να μιλήσω τώρα για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής γνωρίζουμε τις προβληματικές, τα προβληματικά θέματα, τα προβληματικές περιοχές. Ε, πρέπει να περιμένουμε από την Κομισιόν λοιπόν τις νομοθετικές προτάσεις ε, για τη μεταρρύθμιση του βασικού κανονισμού της κοινής, ε, ε, του κοινού οργανισμού αγοράς πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας θα περάσει βέβαια στην αρμοδιότητα της επόμενης προεδρίας στους πολωνούς συναδέλφους. Ένα θέμα της προεδρίας μας λοιπόν είναι το μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ε, διαμορφωθεί από τις κοινέ πολιτικές. Η κοινή πολιτική αλίας είναι... Έχει ένα μέλλον παρόμοιο με την κοινή αγροτική πολιτική να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις ε, κρατώντας τις ίδιες αξίες. Επίσης, θέλουμε ασφάλεια στα αλληλευτικά προϊόντα, υψηλή ποιότητα και βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα λοιπόν για τα προεδρότα της Αλίας ε, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την διατροφική ασφάλεια. Στην κοινή αλληλευτική πολιτική Βέβαια, δεν ασχολούμαστε αποκλειστικά με την αλία. Δεν έχουμε μόνο τρόφιμα με τα οποία ασχολούμαστε. Γιατί ε, ο τομέας της αλίας έχει μεγάλες επιπτώσεις ε, και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και αυτή είναι μία από τις προκλήσεις για την ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η κοινή αλιευτική πολιτική θα συμβάλλει στην ε, διατήρηση του τρόπου ζωής ε, των παράκτιων ε, κοινοτήτων, θα διατηρήσει και θα αυξήσει την απασχόληση και θα βοηθήσει στην αντιμεκών προβλημάτων. Αυτά είναι σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία της κοινή αλληλευτικής πολιτικής που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας καθώς συζητούμε για τη μεταρρύθμιση. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής ηχθειοκαλλιέργειας είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και είναι πολύ σημαντικό να ε, προμηθεύουμε ε, την εσωτερική αγορά με τέτοια προϊόντα. Περιμένουμε τις προτάσεις της Κομισιόν τον Μάιο και μετά θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων ε, στο Συμβούλιο τον Ιούνιο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα και προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας είναι ε, να γίνει πιο ισχυρή η Ευρώπη. Και αυτό είναι μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβουμε ενώπιον των μελλοντικών γενεών. Αυτό ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και αλλιεύματα στο μέλλον, ψάρια. Αλλά και αλλιείς. Αυτό είναι πιο εύκολο να το λέμε παρά να το κάνουμε, γιατί υπάρχουν βραχυπρόθεσμες πιέσεις. Το προηγούμενο μήνα είχαμε ε, τις διαπραγματεύσεις για τα ΤΑΚ και τις ποσοστώσεις, οι οποίες ε, για τα πολυετή, ε, γι' αυτό το λόγο είναι και, ε, αυτό το λόγο είναι και τα πολυετή σχέδια τόσο σημαντικά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν το πολιτικό πρόβλημα, πώς ε, δηλαδή θα πουλήσουμε ε, ε, πώς θα πουλήσουμε στο λαό τις θυσίες της βραχυπρόθεσμες για ένα μακροπρόθεσμο όφελος. Αυτό θα, το πρόβλημα θα επιληθεί ε, θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους. Και μετά με μικρά βήματα θα μπορέσουμε βραχυπρόθεσμα να έχουμε μια ε, αποδεκτή πολιτική οικονομική ε, πολιτική. Γι' αυτό έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα μακροπρόθεσμα σχέδια. Για το Σαβρίδι ε, έχουμε ε, ψηφίσει ένα συμβιβασμό για τον κανόνα ελέγχου της αλίας. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει στο Συμβούλιο και αν μπορεί να μας βοηθήσει. Ε, υπάρχουν φυσικά διαφορετικές απόψεις μέσα στο Συμβούλιο και θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να έχουμε μια κοινή άποψη. Επίσης ε, πρέπει να βρούμε ε, έναν τρόπο να βρούμε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνονται οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα δώσει. Γνωρίζουμε τις απόψεις και ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι το σχέδιο δεν αντικατοπτρίζει τις συνθήκες, ότι πρέπει να ε, αρθεί το σχέδιο αυτό και να ε, δημιουργηθεί ένα καινούριο. Οι φίλοι από την ε, ανατολική πλευρά περιμένουν εδώ και καιρό για τα σχέδια αυτά, τα οποία είναι σημαντικά για αυτούς, ε, γιατί εάν υιοθετηθούν, στην ουσία θα μπορέσουν να πραγματοποιηθεί η προμακροπρόθεσμη εκμετάλλευση όλων των αλλιευμάτων. Το πρόγραμμα... Αυτό λοιπόν είναι ε, σε πρώτο πλάνο θα λέγαμε. Το πελαγικό σχέδιο είναι πολύ σημαντικό γιατί θα είναι το πρώτο σχέδιο το οποίο θα έχει μια πραγματική προσέγγιση οικοσυστήματος. Θα λάβει ε, υπόψη του την αλληλεπίδραση μεταξύ των ειδών του μπακαλιάρου ε, ως ε, θηρευτή και της ρέγκας ε, και της παπαλίνας ως ε, θύραμα. Θα μας επιτρέψουν να δούμε εάν θέλουμε ένα οικοσύστημα το οποίο, στο οποίο θα κυριαρχεί ο μπακαλιάρος ή η παπαλίνα ή μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία. Έτσι λοιπόν ε, τον Απρίλιο πρέπει να γίνει μια πολιτική συζήτηση για τον Βαλτικό Σολομό και τα Βαλτικά Πελαγικά είδη τον Ιούνιο. Επίσης υπάρχουν άλλα τρία θέματα τα οποία θα ήθελα να θίξω ε, τα οποία έχω κληρονομήσει από, τους, ε, από τη Βαλτική Προεδρία. Το καθένα με τον τρόπο του θα βοηθήσει καλύτερα στην εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Το πρώτο θέμα. Μιλάμε για την επιμήκυνση και την παράταση που θα δοθεί σε συγκεκριμένα τεχνικά ε, μέσα, τα οποία ήταν προσωρινά για το Βόρεια Θάλασσα και τον Ατλαντικό, τα οποία λήγουν τον Ιούνιο. Πρέπει γρήγορα να αποφασίσουμε μέχρι τον Μάρτιο το αργότερο, έτσι ώστε να έχουμε χρόνο για υιοθέτηση και δημοσίευση. Ε, εάν δεν γίνει αυτό θα έχουμε κενό νομικό. Νομίζω αν έχω σωστέ πληροφορίες ότι σήμερα συζητιέται αυτή η πρόταση. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την μεταφορά των μέτρων της κοινή αλληλευτικής πολιτικής για την ε, ε, Μεσόγειο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις για το ποια στοιχεία θα πρέπει να αναθέσει κατά εξουσιοδότηση Κομισιόν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ένα τρόπο να συμβιβάσουμε τις απόψεις και να υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Επίσης, ε, παρόλα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολύ συγκεκριμένες απόψεις, έτσι λοιπόν έχουμε λίγο χώρο για χειρισμούς στην Προεδρία. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με την χρηματοδότηση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και την ε, αναθεώρηση του θαλάσσιου δικαίου. Χαίρομαι που βλέπω ότι σήμερα θα ψηφίσετε γι' αυτό και παρόλο ε, και γι' αυτό το λόγο, επειδή η εργασία αυτή είναι ρουτίνα, θα μπορέσουμε γρήγορα να την κλείσουμε. Και τέλος, ε, το βασικό θέμα, ε, με το, οποίο θα, το τελευταίο θέμα μάλλον με το οποίο θα ασχοληθεί η Προεδρία μας, είναι τα δυτικά ύδατα και οι προσπάθειες που γίνονται εκεί. Ε, υπάρχουν δύο πτυχές. Η πρώτη έχει να κάνει με το γενικό σύστημα προσπαθών για τα δυτικά ε, ύδατα που συμφωνήθηκε το 2003. Η Κομισιόν έχει αναθεωρήσει αυτό το σύστημα και τον Απρίλιο θα συζητηθεί ξεκάθαρα το θέμα στο Συμβούλιο. Το, η δεύτερη πτυχή είναι οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τα βενθοπελαγικά είδη. Το 2002 ε, αυτό το θέμα αποκόπηκε από, τις, από το Γενικό Καθεστώς Προσπαθειών για τα Δυτικά Ήβατα και η Κομισιόν τώρα προτείνει μία τροποποίηση του κανονισμού για τα βενθοπλαϊκά είδη. Ε, θα έχουμε λοιπόν μία ε, συζήτηση πολιτικής τον Απρίλιο στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα και για τα εξωτερικά ζητήματα. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα. Έχουμε κάποιες ε, συνθήκες εσωτερικής σχέσης και πρωτόκολλα τα οποία ε, θα πρέπει να ανανεωθούν. Μεταξύ αυτών το πιο σημαντικό είναι το πρωτόκολλο με το Μαρόκο. Από αυτή την άποψη δεν έχουμε ακόμα κάποια πρόταση από την Κομισιόν. Ξέρω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν ε, πολύ παγιωμένες απόψεις για αυτά τα θέματα σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα προτείνει η Κομισιόν. Ένα δεύτερο θέμα είναι η συμφωνία με τη Χιλή για τον Ξηφία. Στην Επιτροπή Αλίας αποφασίστηκε να γίνει ψηφοφορία για αυτό το θέμα. Αυτό έχει πολιτική σημασία. Γιατί θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, όπως καταλαβαίνω. Εμείς στο Συμβούλιο υποστηρίζουμε αυτή τη συμφωνία, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί, καθώς είναι το πρώτο σημαντικό βήμα στη συνεργασία με την Χιλή στον τομέα αυτό. Και στον τομέα αυτό γνωρίζω ότι ως τώρα δεν ήταν δυνατή συνεργασία. Όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, έχουμε μία πολύ βαριά ατζέντα. Ενώ τα μάτια μας θα ε, είναι στραμμένα προς την ε, μεταρρύθμιση της κοινή αλευτικής πολιτικής, ε, δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας ταυτόχρονα και την πρόοδο σε μακροπρόθεσμα σχέδια. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει λειτουργήσει και έχουμε δρέψει τους καρπούς ως τώρα. Επίσης, ε, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δείξουμε στο κοινό ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι ικανά να συνεργαστούν για το συμφέρον του τομέα της αλληλείας ε, και των ε, πολιτών μας. Σας ζητώ λοιπόν την υποστήριξή σας και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Μία ώρα έχει ο Υπουργός στη διάθεσή του. Πρώτος γύρος με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και μετά θα μιλήσουν οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί. Να είστε σύντομοι παρακαλώ για να απαντήσει ο υπουργό. Για το ΕΛΚ, ο κύριος Αντινόρο έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω εκ μέρους του ΕΛΚΑ Η Προεδρία σας αναζωογονεί τις ελπίδες μας διότι όντας μια Προεδρία η οποία είναι μακριά από οποιοδήποτε κέντρο συμφέροντος στον τομέα της αλίας ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να μας βοηθήσει και μας να βρούμε ισορροπημένες λύσεις. Δεν θα κάνω τεχνικές ερωτήσεις, μερικές θεωρήσεις μόνο θέλω να κάνω. Μιλήσατε για λογική διαχείριση της αλίας, για μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, του θαλασσιού που Θέλω να ρωτήσω το εξής. Διαπίστωσα ότι πριν από δεκαετίες οι γεωργοί θεωριόντουσαν οι φτωχοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ οι Ελλείς ήταν οι πλούσιοι. Σε αυτές τις δεκαετίες τα πράγματα άλλαξαν. Φτώχυναν οι ψαράδες και πλούτησαν οι γεωργοί. Πολύ καλό πράγμα για τους γεωργούς. Αλλά δυστυχώς φτώχυνε ο τομέας της αλίας. Μπορεί να μην φταίει και κανείς. Μπορεί να φταίει και ο ίδιος επαγγελματικός ε, κλάδος ο οποίος ε, δεν πρικοδοτήθηκε με ε, νέα μέσα, με κατάρτιση ή δεν βοηθήθηκε από τα θεσμικά όργανα. Να ρωτήσω λοιπόν και σε εσά και στην Κομισιόν. Είναι δυνατόν εμείς να αλλάξουμε το ρόλο του Ευρωπαίου ψαρά και να τον κάνουμε επιχειρηματία. Σε ορισμένες χώρες κάτι τέτοιο έχει επιτευχθεί. Αλλά σε άλλες όχι, διότι πέρα από τις ποσοστώσεις, την αηφόρο, αλληλεία κλπ. πρέπει να διασφαλίσουμε την οικονομία αγοράς σε αυτόν τον τομέα και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να μετατραπούν οι αλληλείς μας σε επιχειρηματίες. Η Ουγγρική Προεδρία που θα προθήσει με σίγουρος λαμπρά τις διακηρύξεις της θα μπορέσει να βάλει τις βάσεις σήμερα ούτως ώστε να γίνει αυτή η μετατροπή. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόδους, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ χαιρετώ τον Υπουργό που βρίσκεται εδώ. Χαίρομαι που μίλησε πολύ για την ε, βιωσιμότητα και αριφορία και θέλει να δουλέψει γι' αυτό και, ότι, και για το γεγονός ότι τα οικονομικά στοιχεία δεν είναι μόνο ε, η προτεραιότητά του, αλλά είναι και η οικολογία. Ε, χαίρομαι επίσης για το γεγονός ότι θέλουμε να συζητήσουμε για την εφαρμογή μακροπρόθεσμων σχεδίων, όπως επίσης χαίρομαι ότι, ε, που είπατε ότι θα εφαρμοστεί η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Τρία είναι τα βασικά θέματα που και εμείς εδώ συζητούμε. Το χρονοδιάγραμμα, τα ζητήματα, ε, όλα αυτά που, που αφορούν στην Αλία, δεν θα τα επαναλάβω, αλλά και η συμμετοχή στην Συμφωνία της Αλίας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πιο αναλυτικά ε, τι πιστεύετε για αυτά. Η παρουσίασή σας ήταν ε, ενδιαφέρουσα, όμως ούτως ή άλλως υπάρχουν ε, στη μερίσια διάταξη κάποιοι στόχοι και θα ήθελα να μας πείτε για τον καθένα από αυτούς ξεχωριστά ως Ουγγρική Προεδρία πώς θα τους αντιμετωπίσετε. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο ε, πρέπει να αποφασίζει από κοινού και η συζήτηση ε, δεν είναι πάντα εύκολη. Είναι γνωστό όμως εσείς είστε αυτοί που θα καθοδηγήσετε τη συζήτηση, θα δώσετε κάποιες ιδέες και θέλουμε να δούμε πώς αυτές οι ιδέες θα μπορέσουν να γίνουν πράξη από την Ουγγρική Προεδρία. Αυτά που μας είπατε δεν αρκούν. Ίσως ε, αν δεν μπορείτε να μας τα αναλύσετε όλα εδώ, μπορείτε και γραπτός να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλαχερ για τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπως και οι συνάδελφοί μου και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Υπουργό που ε, προεδρεύει αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι, χαίρομαι. Που, ε, μια χώρα η οποία δεν είναι ιδιαίτερα, μια χώρα που διαθέτει θάλασσα, αναλαμβάνει την Προεδρία ωστόσο ε, ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει και κοινωνική διάσταση. Είπατε ότι στους προσεχείς έξι μήνες θα αφήσετε τη δική σας σφραγίδα σε αυτόν τον τομέα. Βεβαίως, ε, ε, θέμα είναι η αηφορία. Η αηφορία ενδιαφέρει το Συμβούλιο αλλά και εμάς, το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν. Και βεβαίως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ο ίδιος ο κλάδος, ο τομέας. Και ο ίδιος ο κλάδος ε, κάποια στιγμή έδωσε την εντύπωση ότι απομακρύνεται από την έννοια της αηφορίας. Ωστόσο, ό,τι γίνεται θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την αηφορία. Βεβαίως, εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες. Εμείς είμαστε αυτοί που θα φροντίσουμε αυτόν τον κλάδο με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και δίδεται έμφαση στα μέτρα ελέγχου. Και τούτο θα συμβάλλει στην ανανέωση πολλών αποθεμάτων. Ε, βεβαίως πάντα αναζητούνται συμβιβασμοί. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία και εγώ ως εισηγητής εντυπωσιάστηκα στη, συνεδρίαση του, στη συνάντηση του Συμβουλίου μαζί μου. Ε, δυστυχώς όμως τώρα η κατάσταση είναι απογοητευτική. Θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος και με περαιτέρω διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είπατε ότι, ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει τη συμφωνία με τη Χιλή. Η Επιτροπή αυτή είχε, ψήφισε μια θέση 15 προς 5, δηλαδή με συντηρητική πλειοψηφία 3 προς 1 για απόρριψη αυτής της συμφωνίας, υπέρ της απόρριψης και είχαμε λόγους γι' αυτό. Και σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μια συνάντηση με τους χιλιανούς. Σημειώθηκε πρόοδος βέβαια, αλλά εμείς ε, Ήμασταν στο σκοτάδι, δεν ε, ξέραμε τίποτα. Όταν λέμε χιλί ουσιαστικά μιλάμε για ξηφίες και μιλάμε για τον Ισπανικό στόλο. Υπάρχουν όμως και όλα τα πελαγικά ψάρια. Κοιτάξτε το χάρτη της Νότιας Αμερικής και το μήκος της χιλής από το βορρά προς νότον. Αν λοιπόν εικάσουμε ότι τα σκάφη αυτά αλλιεύουν κάπου στο κέντρο, στη δυτική ακτή, Ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση αυτή. Υπήρξε κάποια πρόοδος, βέβαια, αλλά πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία, διότι εμείς έχουμε ε, μεγάλη ευθύνη να μεριμνήσουμε τον κλάδο αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα πραγματικά να σημειωθεί πρόοδος από αυτό. Αν λοιπόν έχετε την ευκαιρία πριν ολοκληρώσετε ε, τις απαντήσεις που θα μας δώσετε, παρακαλώ πείτε μας αν υπάρχουν συγκεκριμένες απόψεις όσον αφορά την περιφερειοποίηση. Ίσως το θέμα απασχολήσει την Πολωνική Προεδρία κατά το δεύτερο εξάμενο αυτού του έτους, αλλά η περιφερειοποίηση είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόεβιν για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Φαζάκα στην Επιτροπή μας εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων. Με χαρά άκουσα τις προτεραιότητές σας κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Συμφωνώ απολύτως ότι είναι πλεονέκτημα να βλέπει κανείς τα πράγματα έξωθεν όταν ηγείται της Ευρώπης και ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή πολιτικής αλίας. Και πράγματι ο στόχος είναι να γίνει σωστή αξιολόγηση και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Ε, η επιλογή των ε, ορθών προτεραιοτήτων είναι ένα σημαντικό θέμα και βεβαίως η αεφορία είναι το πρώτο εξ αυτών, πολύ σημαντικό για τις μελλοντικές γενιές. πρέπει όλοι να παραδεχθούμε ότι ο πλανήτης καλύπτει κατά 72% από ωκεανούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη, δύναμη στον κόσμο. Άρα λοιπόν ε, μας απασχολούν και οι στόλοι μας οι οποίοι αλλιεύουν σε μεγάλες αποστάσεις και το 70% των ηχθείων που καταναλώνονται στην Ευρώπη προέρχονται από ύδατα εκτός Ευρώπης. Η Ευρώπη λοιπόν έχει ευθύνη για το πώς αλλιεύονται τα ψάρια σε ολόκληρο τον ε, πλανήτη. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τόσο τη δική μας αλλιευτική πολιτική όσο και τη θέση μας στα διεθνή φόρα για τις πολιτικές αλληλείας, για να καταποτελήσουμε την παράνομη αλληλεία στο ολόκληρο τον κόσμο και να στηρίξουμε την βιώσιμη αλληλεία και για υπέρ της ανάπτυξης διεθνών σχέσεων για υπεύθυνη αλληλεία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Συμφωνώ επίσης ότι η προσέγγιση από τη σκοπιά του οικοσυστήματος είναι ορθή προσέγγιση που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κοινή πολιτική αλίας. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα είναι πιο συγκεκριμένα παραδείγματα των προτεραιοτήτων της Ουγγρικής Προεδρίας. Θα οργανώσετε κάποιες διασκέψεις, θα αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες και ποιες ως προς την αηφορία παραδείγματος χάρη. Θα Έχετε ε, κάποιες συγκεκριμένες θέσεις ε, όσον αφορά την παρέτηση από κάποιες ε, περιοχές ή σε σχέση με ενιαίες πολιτικές αλίες. Και η αναθεώρηση της κοινή πολιτικής αλίας μας δίνει μια τεράστια ευκαιρία. Από τη σκοπιά του Κοινοβουλίου η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα στη σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε το δικαίωμα συναπόφαση για τις συμφωνίες που συνάπτονται με ε, τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Και ωστόσο έχουμε λιγότερες πληροφορίες από αυτόν και ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιολόγηση αυτών των συμφωνιών. Ποια είναι η θέση της Ουγγρικής Προεδρίας. Και τέλος, θεωρώ ότι η πολιτική αλίας είναι πάρα πολύ σημαντική και άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον. Πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργού Αλίας, του Υπουργού Γεωργίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος. Υπάρχει συνεργασία με τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Ουγγαρίας επ' αυτού του θέματος. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, διότι αλλιώ ο Υπουργό δεν θα μπορέσει να απαντήσει σε όλου. Ο κύριος Ντρόβατσικ, εκ μέρου του ΕΦΕΧ. Κύριε Υπουργέ, και εγώ σας καλωσορίζω σήμερα εδώ στη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Κατά την εισήγησή σας, κύριε Υπουργέ, επισήρατε την προσοχή μας σε διάφορες πτυχές των προκλήσεων που συνδέονται με την αλία. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αναφερθήκατε στην κοινή πολιτική αλία, στην ανάγκη περαιτέρω δράσης και μεταρρυθμίσεων. Ναι, συμφωνώ. Είναι υψής της σημασίας. Μιλήσατε επίσης για τα πολυετή προγράμματα Αναφέρατε τη Βαλτική. Ελπίζω ότι αυτή θα είναι μια σημαντική πτυχή του έργου σας, δηλαδή το μέλλον της Βαλτικής θάλασσας. Επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στο πλαίσιο αυτό το όλο θέμα το όλο θέμα της αλίας αυτές τις ε, περιοχές. Η γεωγραφική ουδετερότητα στην οποία αναφερθήκατε είναι ε, πράγματι χρήσιμη, συμφωνώ. Πολλές χώρες ε, έχουν άμεσα συμφέροντα όταν αναλαμβάνουν την Προεδρία, άλλες όχι. Ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια ε, περιφερειακή πολιτική και το ε, θέμα της περιφερειοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ε, κύριος Φερέιρα εκ μέρους της Γουέ για τον πρώτο γύρο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Εσείς μιλήσατε για το περιβάλλον, για τις κοινωνικές πτυχές και τις οικονομικές πτυχές. Εγώ θέλω να σταθώ στις δύο τελευταίες πτυχές, την οικονομική και την κοινωνική. Αναφέρατε την τεράστια κρίση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος. Η κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της αλίας δεν έχει ακόμη προσεγγίσει τους βασικούς στόχους. Να εγγυθούμε τη σταθερότητα των αγορών για τα προϊόντα της αλίας και την εγγύηση ενός δίκαιου εισοδήματος για τους αλίες. Οι δύο μεταρρυθμίσεις δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους. Χρειάζεται λοιπόν μία τρίτη η οποία έχει καθυστερήσει, διότι έχει αναβάλει η Κομισιόν την αναθεώρηση της ΚΟΑ και ο τομέας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα σε επίπεδο εσόδων και ανταγωνιστικότητας. Έχουμε επίσης και μία ανισόρροπη κατανομή της προστιθέμενης αξίας μέσα στην όλη αλυσίδα του τομέα. Αν η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες φαίνεται να είναι ανεπαρκείς διότι η μέση δαπάνη την τελευταία δεκαετία ισοδυναμούσε με το μισό των χορηγήσεων της προηγούμενης δεκαετίας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχουμε πρωτοβουλίες εκ μέρους της Κομισιόν, τι μέτρα πρέπει να αναλάβει το Συμβούλιο και τι μέτρα θα αναλάβει η Προεδρία ούτως ώστε να ασκηθεί πίεση για την έγκριση μέτρων που θα εγγυώνται ένα δίκαιο εισόδημα στην αγορά για να αυξήσουν και την προστιθέμενη αξία. Και ρωτώ επίσης την Προεδρία, εσείς ε, δίνετε ιδιαίτερη σημασία στις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Όπως σίγουρα θα γνωρίζετε έγινε μια μεγάλη συζήτηση και σε αυτήν την Επιτροπή για τα πραγματικά αποτελέσματα των τωρινών συμφωνιών συνεργασίας στον αλληλευτικό τομέα. Και ε, εκφράστηκαν τεράστιες αμφιβολίες για την πραγματική για το κατά πόσο μάλλον επωφελήθηκαν οι χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει τις συμφωνίες. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια και υπάρχει και το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Είναι ένα πρόβλημα που το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές. Το να αποκλείσουμε τα νερά της, τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας από τη συμφωνία με το Μαρόκο στον τομέα της Αλίας θέλω να μου απαντήσετε. Κύριε Υπουργέ, με αυτά εμείς τελειώσαμε τον πρώτο γύρο των συντονιστών, των πολιτικών ομάδων και σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Μετά θα μιλήσουν οι υπόλοιποι βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σημαντικά που ετέθησαν και είμαι επεπισμένος ότι τα ζητήματα αυτά θα με βοηθήσουν και εμένα προσωπικά και όλους μας ε, για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που προβάλλουν ενώπιόν μας. Θεωρώ ότι για να είναι επιτυχημένη μια προεδρία πρέπει να γίνει σωστή συλλογή πληροφοριών. Υπάρχουν ε, κάποια κινητά μέσα στην αίθουσα και εμποδίζουν τους διερμηνείς. Ελπίζω ότι σε συνεργασία μαζί σας θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα θέματα. Για την βιωσιμότητα και την αηφορία να πω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη του τομέα. Αν δεν βρούμε κάποια λύση για τη βιώσιμη αλία δεν θα υπάρχουν πλέον αλίες ούτε και αλλιεύματα ούτε και αλία. Η αλία στα εσωτερικά είδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρή σε κλίμακα. Όμως ε, πρέπει να την προσέξουμε γιατί υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες και είναι και πολλοί οι στα παγκόσμια ύδατα που ε, δεν ε, ασκούν την αλληλεία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και βιώσιμο. Τώρα, ε, για τις, αναφέρθηκαν οι ποσοστώσεις. Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Πώς δηλαδή μακροπρόθεσμα θα μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα που θα διατηρήσει τα αλλιεύματα. Ναι, όντως ε, είπατε ότι οι γεωργοί έγιναν πλούσιοι και αλληλείς φτωχοί. Δεν ξέρω οι γεωργοί αν το θεωρούν αυτό. Εγώ ως υπουργό υπεύθυνο για την γεωργία και την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου και την αλληλεία θα πρέπει να έχω μια ισορροπία μεταξύ αυτών των τομέων. Ο καθένας παλεύει για τα δικά του δικαιώματα και πραγματικά οι μάχες δεν βοηθούν. Πρέπει να βρούμε μία ε, λύση η οποία θα κρατήσει σταθερό τον κλάδο. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι η κοινή αλλιευτική πολιτική μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ε, μιλάμε για παραμέληση ή για αναβολή. Ε, εδώ ουσιαστικά προσπαθήσαμε να δούμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του 2002. Υπήρχαν πέντε ε, σημαντικά ζητήματα, ε, οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις, το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες, δεν υπήρχε πειθαρχία, ε, γενικά αυτή η αδυναμία ήταν από τα, μέσα στα ζητήματα αυτά. Τον Δεκέμβριο του 2009 θα κλείσει η πρώτη φάση διαβούλευσης και θα βγουν και τα αποτελέσματα της συζήτησης σε ένα έγγραφο τον Απρίλ. Ε, μάλλον έγιναν τον Απρίλιο του 2010 και έκτοτε έγιναν θεματικά σεμινάρια ε, μια, ένα μεγάλο συνέδριο. Το Νοέμβριο του 2010 έγινε το τελευταίο συνέδριο, τελευταία διάσκεψη σε σχέση με την μεταρρύθμιση της αλίας. Εκεί αναφέρθηκαν πρακτικές και καινοτόμα σχέδια. Και αυτά θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται η νομοθεσία και τον Μάιο. Περίπου στο τέλος της Προεδρίας υπολογίζουμε να έχουμε αυτό το έγγραφο, δηλαδή μια σύνοψη των εργασιών έως τώρα. Το θεωρούμε σημαντικό να έχουμε ένα πακέτο μεταρρύθμισης ε, εγκαίρως για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε λογικά. Έτσι λοιπόν συνεργαζόμαστε συνεχώς με τους εκπροσώπους της Κομισιόν και προσέχουμε αυτό το σημαντικό έγγραφο. Το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας. Η βιωσιμότητα έχει γίνει μια λέξη κλειδί για την κοινή αλλιευτική πολιτική. Ε, και έχει να κάνει και με το θέμα των παρεμπιπτών των ελιευμάτων τα οποία είναι υπερβολικά και πλητούν και την παραγωγικότητα. Ε, έχει να κάνει με την επιλεκτικότητα των διχτυών, αλλά ε, η πρακτική είναι αυτή που δεν αρκεί, που δεν επαρκεί σχετικά με το πώς θα λύσουμε αυτό το θέμα. και ουσιαστικά τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα δεν ε, πετιώνται και πάλι στη θάλασσα. Το θέμα είναι πόσα είναι αυτά τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα. 8% λέγανε ως τώρα. Μισό εκατομμύριο τόνοι ε, θα μπορούσε να είναι το κατώτατο όριο, αλλά γενικά ε, το θέμα αυτό θα έλεγα ότι είναι προβληματικό και πρέπει να επιληθεί. Και θα πρέπει να το εντάξουμε και στις συζητήσεις της μεταρρύθμισης. Δεν μπορούμε βέβαια να φτάσουμε στο μηδέν, όμως τουλάχιστον να υπάρχει καλύτερη τήρηση των κανόνων. Να εξετάσουμε τους κανόνες ε, για τα δίχτυα να τους ε, αναθεωρήσουμε ενδεχομένως ε, και γενικά να δούμε πώς θα μπορέσουμε να σταματήσει αυτή η κακή πρακτική η οποία είναι πραγματικά ε, μία σπατάλη θα έλεγα και είναι και μόλυνση καθώς πετώνται πίσω νεκρά ψάρια. Θα υπάρξει μια διάσκεψη γι' αυτό η οποία θα είναι και ένα καλό φόρουμ για μια τέτοια συζήτηση. Υπάρχουν επίσης και άλλες ερωτήσεις που θέσατε για να δω ποια θα απαντήσω πρώτη για την ε, Συμφωνία Συνεργασίας με το Μαρόκο. Η συμφωνία αυτή είναι ένα πολύ επίκαιρο και σημαντικό ε, θέμα για το 2011 ε, καθώς θα λήξει το πρωτόκολλο και περιμένουμε τις προτάσεις της Κομισιόν για αυτό το θέμα. Από τη μία λοιπόν η Προεδρία πρέπει να δει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία για μας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε πάντοτε να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν βρισκόμαστε σε θέση διαπραγματευτική. Είμαι πεπισμένος ότι και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εξετάσει και αντιμετωπίσει αυτό το θέμα ε, όσον αφορά για παράδειγμα την εξάντληση των ε, φυσικών πόρων και υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια αποτελέσματα από τις έρευνες των Ηνωμένων Εθνών και είναι το θέμα αυτό μέσα στα, στην ημερήσια διάταξη της διάσκεψης, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ακόμα προτάσεις για το θέμα. Για την συχθειοκαλλιέργειες τώρα, πολλοί θεωρούν ότι οι χθειοκαλλιέργειες αποτελούν λύση για το πρόβλημα της αλίας. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλές ε, βέβαια αντικρώμενες απόψεις και υπάρχουν και κράτη που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Απ' την άλλη υπάρχουν ε, διαφωνίες σχετικά με το πόσο ε, ανθυρή οικονομικά μπορεί να είναι η χθιοκαλλιέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε πάρει τη σωστή κατεύθυνση όταν λέμε ότι οι χθιοκαλλιέργειες πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο ειδικότερα σε επίπεδο επιστημονικών ερευνών. Είμαι πεπισμένος ότι ο τομέας αυτός πρέπει απαραίτητα να ε, αναπτυχθεί στην Ευρώπη. Από την άλλη όμως πρέπει οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε να είναι περιβαλλοντικά φιλικές και να εξετάζουμε τις ηχθειοκαλλιέργειες σε, ε, σε συνδυασμό με άλλους, άλλες πολιτικές. Να δούμε πώς η συνεργασία με τις τρίτες χώρες μπορεί να περπατήσει και να φροντίσουμε να τηρούνται οι κτηνιατρικοί κανόνες. Όσον αφορά την υγεία των ε, ζώων και των ε, ψαριών, θεωρούμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά προϊόντα υψηλού επίπεδου, τα οποία έχουν την αγορά τους και οι πολίτες δεν θέλουν να ρισκάρουν να μην έχουν υγιή ψάρια, ακόμα και αν αυτά είναι από ηχθειοκαλλιέργειες. Συνεχώς λοιπόν ενημερώνονται σχετικά με τη σήμανση των ε, αλλιευμάτων και η σήμανση είναι κάτι που ενδιαφέρει τους πολίτες, όπως και η βιώσιμη ηχθειοκαλλιέργεια. Και μέσα στον τομέα της αλίας οι χθεοκαλλιέργειες έχουν αυξηθεί. Αυτό είναι πραγματικά ένα ξεκάθαρο σημάδι του πού πηγαίνει το πράγμα. Τώρα για τα μακροπρόθεσμα σχέδια, για ο γάβρο, για παράδειγμα. Εδώ υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις. Εγώ στην, απάντηση, μου έχω ήδη εκφράσει την άποψή μου. Ε, είμαι κάπως ε, αισιόδοξο, γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξει συμφωνία. Το Κοινοβούλιο έχει πίσω του την πρώτη ανάγνωση και για τα δύο σχέδια. Τώρα χρειαζόμαστε μια κοινή θέση. Και ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα μπορούσε με αυτό το γνώμα να συνεχίσει. Θα κάνω τα πάντα λοιπόν για να είναι επιτυχημένος αυτός ο διάλογος και να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε και ελπίζω ότι θα προχωρήσει το θέμα και στο Συμβούλιο. Τώρα για το Γάβρο ε, υπάρχει μια, ένα σχέδιο ε, το οποίο δεν ε, συνάδει με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το Γάβρο. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε το, το έγγραφο της Κομισιόν ε, για να μπορέσει να συζητήσει το Συμβούλιο τα σχέδια και όταν έχουμε αυτές τις προτάσεις τον Απρίλιο και τον Ιούνιο θα έχουμε συζήτηση στο Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. Μέσα στα πλαίσια της ε, νέας κοινή αλληλευτικής πολιτικής λοιπόν θα πρέπει να επιληθούν αυτά τα ε, θέματα. Τώρα για το, η συμφωνία για τον Ξηφία με τη Χιλή. Αναφέρθηκε και αυτό στις 3 Ιουνίου. Υπερψήφισε την συμφωνία ε, το Συμβούλιο σχετικά με τα λιεύματα Ξηφίας στον ε, Ειρηνικό οι υπηρεσίε του Συμβουλίου είναι σε επαφή με τη Χιλή για την υπογραφή και η υπογραφή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, μία ε, πρώτη εφαρμογή, όμως η Επιτροπή Αλίας δεν έχει υποστηρίξει την υπογραφή. Αυτό φυσικά είναι δυνατόν, στην Ολομέλεια δηλαδή, να υπάρξει μια άλλη άποψη γιατί θεωρώ πως ε, είναι λυπηρό εφόσον τα κράτη-μέλη έχουν υποστηρίξει τα αποτελέσματα της ε, συμφωνίας, τα, τα συμπεράσματα συγγνώμη, της συμφωνίας. Κάποια άλλα θέματα τώρα που αναφέρατε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό στα διαφορετικά περιφερειακά συστήματα να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου, Κομισιών και Κοινοβουλίου. Εγώ προσωπικά έχω ενημερωθεί σχετικά με, την Βορεια... με τη Βαλτική και θεωρώ ότι σχετικά με το σολομό στη Βαλτική και άλλα είδη θα μπορέσουμε να έχουμε τα ε, επιθυμητά αποτελέσματα. Τέλος. Να μιλήσω για τις δυνατότητες που έχουμε για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιτυχημένη όταν ε, μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά τα διάφορα θεσμικά ε, όργανα μεταξύ τους, όταν ε, επιλύονται τα προβλήματα. Αυτή η διαθεσμική συνεργασία λοιπόν είναι μια, ένα κεντρικό ζήτημα. Δεν πρέπει ο καθένας να δρά μεμονωμένα, πρέπει να βρίσκουμε από κοινού μακροπρόθεσμες λύσεις. Χρειαζόμαστε μία οριζόντια συμφωνία θα έλεγα έτσι ώστε να είναι αποδεκτές οι λύσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεν, όταν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, θα πρέπει να επιλύουμε τα ζητήματα κατά περίπτωση. Και θα πρέπει να προσέξουμε να ε, πάντοτε να δρούμε με βάση την συνθήκη της Λισαβάνας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Να τελειώσουμε τώρα με τον τελευταίο γύρο των τοποθετήσεων. Διαβάζω τον κατάλογο των ομιλητών. Ωραία. Η κυρία Δελμπαρέα θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε εσείς για τους κοινούς στόχους για την κοινή πολιτική αλληλείας, για τις επιστημονικές βάσεις που αποτελούν και το θεμέλιο της κοινή πολιτικής, μιλήσατε για χρηματοδότηση και κοινωνικό χαρακτήρα. Ρωτώ, τι ρόλο θα παίξει αυτή η Προεδρία για την απαράκτια αλία και για το ρόλο της γυναίκας στον τομέα της αλίας. Εσείς ε, μιλήσατε για τις ε, δυσκολίες συμφωνίας που έχουμε και με τις εντεταλμένες πράξεις ε, πώς θα το ξεπεράσουμε εμείς αυτό το πρόγραμμα και τα διάφορα είδη πώς θα προστατευθούν με το πρόβλημα ας πούμε με τα σαφρίδια που έχουμε εμείς ε, με το Μαρόκο και με τη συμφωνία του Μαρόκου τι θα κάνετε, πώς θα δείτε εσείς τη νέα μορφή διαχείρισης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, χαίρομαι που μας δώσατε λεπτομερείς απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Και ιδιαίτερως αναφερθήκατε στις απορρίψεις ε, και αναφερθήκατε σε τεχνικά θέματα, ε, επιλεκτικότητα, δίκτυα κλπ. Αυτά βεβαίως δεν είναι μόνο τεχνικά μέτρα, αλλά βασίζονται ε, και σε συγκεκριμένα μέτρα. Το κοινό όμως ε, μπορεί να περιμένει για να δει πότε εμείς θα αποφασίσουμε την μεταρρύθμιση της κοινή πολιτικής αλίας και όταν το 80% των αποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα γίνονται αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης και ε, συνεχώς βλάπτουμε τα θαλάσσια αποθέματα. Τι θα απάντησε θα δώσει η Ουγγρική Προεδρία προς το κοινό. Το κοινό το οποίο μας κατακλείζει με τηλεφωνήματα και μηνύματα στα μέλη αυτής της Επιτροπής. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που θα λάβετε για να διασφαλίσετε ότι τα θα δοθεί τέλος της απορρίψης των παρεμπιπτών των αλλιευμάτων. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό και να ευχηθώ στην Ουγγλική Προεδρία κάθε επιτυχία. Έχω την εξή ερώτηση, είναι πολιτικής φύσεως. Ο Υπουργό ε, αναφέρθηκε στο Μαρόκο και είπε ότι ελπίζει ότι η Κομισιόν θα υποβάλει μια πρόταση. Ωστόσο η απάντηση που εγώ περίμενα ήταν η εξή. Εγώ θα ήθελα να μάθω πώς η Προεδρία βλέπει αυτό το θέμα από πολιτική σκοπιά. Δηλαδή το θέμα με το Μαρόκο είναι σύνθετο. Έχει και πολιτικό περιεχόμενο. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει πολιτική σταθερότητα στη Βόρεια Αφρική για την Ευρώπη και το παράδειγμα της Τινησίας είναι απολύτως ξεκάθαρο. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν για τα αλλιευτικά θα λάβουν υπόψη τους διμερείς, τα διμερείς συμφέροντα και ακόμα και τα πολιτικά. Θέλω λοιπόν να ξέρω αν θα σημειωθεί η πρόοδος στο ξεμπλοκάρισμα αυτού του ζητήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας ε, χαιρετήσω και χαίρομαι που μπορέσαμε να έχουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε. Αναφέρεται ότι ε, στην Αλία μια ανοιχτή θάλασσα ε, σε μια ανοιχτή θάλασσα πρέπει να ληφθεί υπόψη το οικοσύστημα και η ανταλλαγή των ειδών. Εγώ έχω να μιλήσω για το θάνατο των ε, αλλιευμάτων, το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό. Είναι και θέμα του οικοσυστήματος. τουλάχιστον για τα εσωτερικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κομμάτι της αλίας μας, ε, ελπίζω ότι στην νομοθεσία θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή γιατί είναι σημαντικό να δούμε και αυτό το ζήτημα. Τώρα για τις ηχθειοκαλλιέργειες που είναι όχι μόνο στην ανοιχτή θάλασσα αλλά και σε κλειστά συστήματα και αυτό θα ε, έδινε τη δυνατότητα σε πολλά ε, κράτη που δεν έχουν θάλασσα να αναπτύξουν ηχθειοκαλλιέργειες και να ε, παράγουν ψάρια. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, για, κύριε Υπουργέ συγγνώμη, για τις ερωτήσεις σας, για τις απαντήσεις σας. Να σας ρωτήσω για τις αντσούγες. Εσείς ε, μας μιλήσατε για καλή θέληση και ρωτώ. Έτσι όπως μας έρχεται η πληροφόρηση, το Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να αποσύρει το σχέδιο. Κατά δεύτερο, για τα τον αλλιευτικά που εργάζονται ε, στον Ινδικό έχουν πρόβλημα με την πυρετία. Δεν είναι βέβαια μόνο τα αλλιευτικά που υποφέρουν, αλλά εμείς ε, είχαμε ένα ψήφισμα να συμπεριληφθούν και τα αλλιευτικά στη Συμφωνία Ατλάντα, διότι είναι και τα πιο ε, αδύναμα να προστατευτούν πλοία. Λοιπόν, τι σκοπεύετε να κάνετε για να βελτιώσετε την ασφάλεια των, των αλλιευτικών που ψαρεύουν στον Ινδικό. Έχουμε και μία απόφαση της 14ης Ιανουαρίου του 2011 για μερικά μέτρα στην ακτή του Ελεφαντόδοντος ε, για το θέμα της μη μεταφοράς κονδυλίων. Και υπάρχει ένας ισπανικός κλάδος που δεν μπορεί να προσεγγίσει το λιμάνι του Αμπιτζάν. Δεν είναι όμως μόνο πρόβλημα των ισπανικών αλλιευτικών. Είναι και ο κόσμος ο οποίος ζει με τα ισπανικά αλλιευτικά τα οποία καταπλέουν στο λιμάνι. Ρωτώ λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε κάτι σχετικά. Τι λύσεις έχετε κατά νου για το μέλλον. Κύριος Μιλάνα. Grazie. Grazie signor Ministro. No, due sole considerazioni. Mm, io credo che lei abbia molto chiaro la vicenda. Είναι σαφές ε, το θέμα της αλίας ε, στο Μαρόκο. Υπάρχουν και χιλιάδες ανθρώπινες μοίρες που συνδέονται με όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει λοιπόν εμείς να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα το οποίο ξεπερνάει τα όρια της ε, πολιτικής και το θέμα της ε, Δυτικής Σαχάρας είναι μία μεγάλη ιστορία και πρώτα όσο νωρίτερα αναλυθούν πρωτοβουλίες τόσο το καλύτερο. Τώρα, πριν από έξι μήνες το Κοινοβούλιο ψήφισε μία γνωμοδότηση αρκετά πλήρη και ζητούσε να υπάρξουν ρυθμίσεις για το θέμα. Ρωτώ, είναι και η ώρα για κάτι τέτοιο, δεσμεύεται η Προεδρία να το πράξει είναι ένας τομέας που δεν αφορά μόνο τη θάλασσα αλλά και άλλα γενικότερα πολιτικά ζητήματα. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις τοποθετήσεις, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που θέσατε τόσες πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσες περισσότερες γίνεται. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να μιλάμε για το ρόλο των γυναικών. Πρέπει να προσέξουμε ώστε οι γυναίκες ε, να την χάνουν της κατάλληλης προσοχής ε, σε αυτόν τον δύσκολο κλάδο. Θεωρώ ότι η συζήτηση για αυτό το θέμα ε, είναι πολύ μεγάλη για να μπορέσει να βελτιωθεί ο ρόλος των γυναικών. Πολλά ζητήματα Επίσης, πολλές ερωτήσεις ε, ε, τέθησαν για την ε, συμφωνία με το Μαρόκο. Είναι τα λογικά, τα πολιτικά ζητήματα σχετικά με αυτή την συμφωνία. Είναι μεγάλη ιστορία με την Δυτική Σαχάρα, το Μαρόκο και αυτά τα ύδατα είναι μια περιοχή κρίσης, η περιοχή της Βόρειας Αυτηρικής και υπάρχουν διάφορες απόψεις στο Συμβούλιο σχετικά με τη λύση των ζητημάτων που αφορούν στην περιοχή αυτή. με την κυρία Επίτροπο αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή και εξετάζουμε τη λύση. Ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Η Μαυριτανία είναι άλλος ένας, άλλη μια περιοχή ε, που είναι πολύ σημαντική και υπάρχει μια συμφωνία με τη Μαυριτανία. Υπάρχουν ευαίσθητα ε, ζητήματα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ειδικότερα όταν μιλάμε για συμβιβασμό. Πρέπει να ε, συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει και ανταγωνισμός για τις απορρίψεις ηχθείων και τι πρέπει να περιμένουμε για από το 2013. Η αλληλευτική πολιτική θεωρείται ότι θα λειτουργεί ως έχει μέχρι το 2013. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις, ε, όμως ο τομέας της ε, αλληλείας πρέπει να εξετάσει λύσεις για το πώς θα, μειωθούν οι απορρίψεις. Υπάρχουν είδη που δεν είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και μάλιστα πολλά από αυτά είναι προστατευόμενα και αυτά απορρίπτονται ως τα λιεύματα στη θάλασσα. Τώρα για τα λιεύματα στα εσωτερικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χαίρομαι που θέσατε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα τομέα ε, που εμπίπτει στην εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Υπάρχουν εθνικοί σχετικοί κανονισμοί, νομοθεσίες για τα εσωτερικά ύδατα και η κατάσταση είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα. Στην Ουγγαρία είναι παρόμοια η κατάσταση. Και με εθνικούς κανόνες ρυθμίζεται ο αριθμός των αλλιευμάτων που επιτρέπεται σε κάθε περιοχή χώρες που δεν έχουν παράκτιες περιοχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την ηχθειοκαλλιέργεια ως μια νέα δυνατότητα. Θα πρέπει να προσέξουμε τους κλιματικούς παράγοντες και αν το κάνουμε αυτό ε, θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γενικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε ενδελεχώς στο μέλλον. Να διασφαλίσουμε επίσης την κοινή αλλιευτική πολιτική. Τον Ιούνιο του 2011 θα υπάρξει ε, απόφαση του Συμβολίου. Τώρα για την πειρατεία. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές περιοχές ε, στον κόσμο που πλήττονται από αυτό το πρόβλημα. Στο παρελθόν δυστυχώς δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τους πειρατές και να προστατέψουμε παρκώς τα λιεύματα στις περιοχές αυτές. Πρέπει να γίνει πιο λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης και γι' αυτό θα μπορούσα θα μπορούσα να σας στείλω γραπτό στην απάντησή μου, όπως και απάντηση για τα θέματα σχετικά με την ακτή του ελεφαντοστούν. A szardellával kapcsolatban meg tudjuk erősíteni azt, hogy a Σχετικά με το γάβρο, να επιβεβαιώσω ότι η Βελγική Προεδρία ζήτησε από την Κομισιόν να πάρει πίσω την πρότασή της. αγαπητοί βουλευτές, προσπάθησα να απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και την προσοχή σας. Eh, eh, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ήσασταν και γενναιόδωρος του χρόνου που μας αφιερώσατε. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Τις προάλλες ο Πρωθυπουργός σας είπε ότι αυτή η Προεδρία θα είναι φιλική προς το Κοινοβούλιο, το ελπίζω κι εγώ και ελπίζω ότι η συνεργασία θα γίνει σε με τον απόλυτο σεβασμό της Λισαβόνας. Εγώ πάντα αστιευόμενη, πάντα λέω ότι το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο συμφωνεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ η Κομισιόν και το Συμβούλιο πέρα βρέχει. Εγώ προτείνω, εγώ πάντως σας λέω ότι θα είμαστε καλοί συνεργάτες, τουλάχιστον εμείς, Πάντως το μόνο που μπορούμε να πούμε έναντι του Συμβουλίου για το Μαρόκο μία έλλειψη μια προφλεκτική έλλειψη, δηλαδή τελειώνει η συμφωνία και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε επιχειρησιακό, διαχειριστικό επίπεδο δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι σημαντικές αποφάσεις. Θα συζητηθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών. Σίγουρα ξέρουμε ότι υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ της Επιτρόπου μας και προσωπικότητων της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Όλα αυτά όμως πρέπει να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο. Όπως και να έχει πάντως κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και εύχομαι η Προεδρία σας όντας η Προεδρία μιας χώρας η οποία δεν έχει και πολύ αλία ε, ελπίζω ότι θα είστε υπεράνω των μερών και θα μπορέσετε να βοηθήσετε καλύτερα. Πάω να αποχαιρετήσω τον Υπουργό. Λοιπόν, αρχίστε να βάζετε τις καρτούλες στο μηχάνημα για να ψηφίσετε.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 συγκητή είναι ο κύριο Ριβελίνη. Παρακαλώ ησυχία εκεί στο βάθο της αίθουσα. Παρακαλώ. Excuse me. Μπορείτε να πάτε να κουβεντιάσετε εκτός αιθούσης παρακαλώ. Όπως λοιπόν γνωρίζετε αυτό το θέμα είναι με ε, τα τακτική νομοθετική διαδικασία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αποφασίσαμε λοιπόν ο εισηγητής και όλοι οι σκεώδεις ή οι εισηγητές αποφασίσαμε ότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε παραπάνω και θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία σήμερα για να περάσει το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Κύριε Ριβελίνη θέλετε να πείτε κάτι ή να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Ριβελίνη. Να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τις πέντε θεωρήσεις που δεν χρειάζεται να τις ψηφίσουμε και μετά ψηφίζουμε όλο το πρώτο μπλοκ των συμβιβαστικών τροπολογιών. Αρχίζει η ψηφοφορία για όλο αυτό το μπλοκ. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται 19 υπέρ και μία αποχή. Πάμε στο δεύτερο σετ ψηφοφορίας ψηφοφορίας, θα ψηφίσουμε χωριστά, ψηφίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία 21. Πέρα στις ψηφοφορίες, 19 υπέρ 2 κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική αριθμός 26. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 38 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συμβιβαστική 40, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Σαράντα ένα, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19-2. Ψηφίζουμε την 42, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε την νομοθετική πρόταση, έτσι όπως τροποποιήθηκε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ ένας κατά ψηφίζουμε το νομοθετικό σχέδιο. Πέρας της ψηφοφορίας. Είκοσι υπέρ ένας κατά εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ριβελίνη. Και θα το συζητήσουμε λοιπόν το Μάρτιο στην Ολομέλη. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, είναι η, μετα... η αλλαγή του κανονισμού για 861-2006 για το δίκαιο της θαλάσσης ο κύριος Φερέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήδη μπόρεσα να διαβιβάσω στους και ηγητές ε, και στους, ε, στους συναδέλφους και στη γραμματεία μία πρόταση. Θα ήθελα να σας αναφέρω εδώ μία προφορική τροπολογία σχετικά με τις τρο... τροπολογίες 6, 7 και 8 για να μειώσουμε το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% αρχικά εγώ αντιπροτείνω 60%. Υπό την οπτική της απόλυξης έναν συμβιβασμό, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη και όλη τη συζήτηση που είχαμε εδώ στην ομάδα, όπως επίσης λαμβάνοντας υπόψη μας και τις γενικές αρχές οι οποίες, ε, με τις οποίες συμφώνησαν πολλοί συνάδελφοι. Η αρχή λοιπόν είναι να, εφαρμό, να προσαρμόσουμε το θέμα στις νέες συνθήκες, όχι μόνο με το πρόβλημα δηλαδή της διαχείρισης των αλληλευτικών αποθεμάτων, αλλά και με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις νέες αρμοδιότητες που εκχωρεί. Νέο λοιπόν θεσμικό πλαίσιο, νέα πραγματικότητα στον τομέα προτείνουμε μία αύξηση της συγχρηματοδότησης οριζόμενη σε αυτό το επίπεδο. Είμαι σίγουρος ότι με αυτή την πρόταση η Κομισιόν θα έχει κάθε ελευθερία απόφασης, την οποία ήδη βέβαια έχει όταν ορίζει τα ανώτατα πόσα για τη συγχρηματοδότηση. Εμείς εδώ απλώς ε, θέτουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε το 50% συγχρηματοδότησης και να φτάσουμε μέχρι το 60%. Αφορά λοιπόν τις τροπολογίες 6, 7 και 8 όπου δεν θα έχουμε 75% αλλά 60%. Λοιπόν, έχει κανείς αντίρρηση στην προφορική τροπολογία, ουδής. Θέλει η Κομισιόν να μιλήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπα δύο φορές στο παρελθόν τα συζητήσαμε. Αν αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για τη συγκέντρωση στοιχείων, αν αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για ελεγχόμενες δαπάνες, αναφίβολα θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερες προσδοκίες για υψηλότερα ε, ποσοστά συγχρηματοδότησης. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση με αυτόν τον τρόπο θα χρηματοδοτήσουμε λιγότερα projects. Άρα λοιπόν η Κομισιόν δεν είναι έτοιμη να δεχθεί μεγαλύτερο ποσοστό συγχρηματοδότηση ούτε για τη συλλογή δεδομένων ούτε για τον έλεγχο. Κοιτάξτε, δεν εκπλήσουμε, διότι η Κομισιόν και στην προηγούμενη συνεδρίαση αναγνώρισε ότι τούτο δεν θα σημαίνει μείωση στον αριθμό των ε, project, των προγραμμάτων. Τώρα λέει το αντίθετο. Όπως είπα και πριν, η Κομισιόν έχει περιθώριο ε, κινήσεων ακόμα και μπορεί να λειτουργήσει μέχρι τα όρια τα οποία έχουν καθοριστεί με την εμπλοκή των χωρών μελών. Αλλά επειδή μιλούμε για συγκέντρωση δεδομένων και ελέγχου, δεν νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι λογική. Ο καθένα είπε τη γνώμη του, πάμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, 13 του κυρίου Καντέκ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε τη 14 του κυρίου Καντέκ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2 του κυρίου Φερέιρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 3 του κυρίου Φερέιρα. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 15 αποσύρθηκε 4 του κυρίου Φερέιρα πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται 5 του κυρίου Φερέιρα πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται 6 του κυρίου Φερέιρα με την αλλαγή που μας πρότεινε προηγουμένως. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 7 υπέρ και 13 κατά. 7 του κυρίου Φερέρα με την προβλεπόμενη αλλαγή. Πέρας ψηφοφορίας. Ίδιος συσχετισμός δυνάμεων. 8-13 απορρίπτεται. Ο 8 του κυρίου Φερέρα. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13-8. 9 του κυρίου Φερέιρα. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 ψήφοι κατά. Δεκαέξι του κυρίου Καντέκ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. 10 του κυρίου Φερέιρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. 11 του κυρίου Φερέιρα. Πέρας ψηφοφορίας. 13 υπέρ και 8 κατά. Ψηφίζουμε το εκτιμώντας ένα. Το τροπολογία στο εκτιμώντας ένα. του κυρίου Φερέιρα, αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται ομόφωνα. Η νομοθετική πρόταση ούτως τροποποιημένη, αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται ομόφωνα. και ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια. Πάμε στο επόμενο σημείο. Συμφωνία συνεργασίας με τις Κομμαόρες και ο κύριος Καπουλασάντος έχει το λόγο. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ελάχιστα να προσθέσω στα όσα λέει η έκθεση. Δεν αλλάζουν, αλλάζουν και πολλά στα όσα είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση. Μιλούμε για ένα πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής στην περιοχή της Μοζαμβίκης, τρία νησιά, 30.000 ε, άνθρωποι συνολικά εμπλέκονται. Η νέα συμφωνία έχει δύο πτυχές, στις οποίες θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας. Και θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι τούτο για την ανάπτυξη του τομέα της αλληλείας στη χώρα αυτή. Αυξάνονται οι δυνατότητες αλληλείας για τον ευρωπαϊκό στόλο. Με τέτοιες συμφωνίες όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάντοτε το πρόβλημα να περιθωριοποιείται η Επιτροπή Αλίας ακόμα και στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Εσείς, Πρόεδρε, γράψατε στην Κομισιόν από αυτού, μάλιστα πρόσφατα, επισύροντας την προσοχή στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τέτοια μορφής συμφωνίας. Βεβαίως, η συμφωνία αυτή Η συμφωνία αυτό τίθεται σε ισχύ προσωρινά για, ε, για φέτος και απλώς θα ήθελα να επισημάνω αυτά τα οποία σας είπα. Ευχαριστώ. Ναι, ε, ε, ρωτήσω κάτι. Α, Θέλω να υποστηρίξω αυτή τη συμφωνία η οποία θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή αλία με νέες δυνατότητες αλίας. Και θέλω να τονίσω ότι η παράταση αυτού του πρωτοκόλου βασίζεται στις αρχές της υπεύθυνη και αηφόρας αλίας αναλυτικά λέει, αναφέρει τι θα αλλιεύουν τα ευρωπαϊκά αλλιευτικά και αποκλείει την εξάντληση των αλλιευτικών πόρων. Να τονίσω ότι 33.000 θέσεις απασχόλησης ε, ε, συνδέονται με την αλληλεία στα νησιά ε, των Κομορών και από αυτές τις 33.000 θέσεις μόνο 16.000 έχουν να κάνουν με την τοπική αλία με αυτήν τη συμφωνία αυξάνονται οι επενδυτικές δυνατότητες στον τομέα της αλλήλεια, αλλά αυξάνονται και δυνατότητες απασχόλησης. Είναι σαφέστατο επίσης στις συμφωνίες τι είδους αλλιευτικά ψαρεύουν στην περιοχή. Και ελπίζουμε ότι με την επιστολή που έχει στείλει η Πρόεδρος θα βελτιωθούν και οι σχέσεις της Κομισιόν με το Κοινοβούλιο. Πρέπει να είμαστε απαιτητικοί προς την Κομισιόν ζητώντας διαφάνεια νομιμό και νομιμότητα διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος ε, για να ε, εμφυσίσουμε ε, πνοή στην συμφωνή, στη συνθήκη της Λισαβόνας Α, η κυρία Λέβιν, τελευταία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Την ε, αξιολόγηση που μπορέσαμε εμείς να λάβουμε, που είναι απλώς μια σύντομη έκθεση, δεν είναι το σύνολο της έκθεσης, είναι μια περίληψη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδεχθούμε. Διαρωτώ με, ο εισηγητής έχει την πλήρη αξιολόγηση ή όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο θα έπρεπε να έχει πρόσβαση ολόκληρη η Επιτροπή και θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για κάτι το οποίο βλέπω εγώ σε αυτή την ε, σύνοψη και εκεί και αφορά την υπερεκμετάλλευση των ηχθιδίων, των γόνων και εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία με τις αρχές των Κομορών για τη βελτίωση των συνθήκων αλίας. Αυτό ήθελα να πω. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο θα μιλήσω εγώ. Λοιπόν, αύριο θα κάνω, τα, θα κάνω και τα σχετικά σχόλια με την απάντηση που μου στείλει η κυρία Δαμανάκη. Εγώ ε, διερευνώ τι γίνεται με την ε, έκθεση αξιολόγησης εξπόστε και όταν θα έρθει η Επίτροπος την πρώτη του μηνός θα της ε, πούμε ποια είναι η θέση μας σοβαρά. Αύριο θα σας πω τι γίνεται με τη διαθεσμική συμφωνία που θα έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο ανταλλαγής πληροφόρησης που ισχύει μέχρι σήμερα. Η, απάντηση που, η ερώτηση που κάνατε εσείς στον, που στον Υπουργό και δεν σας απάντησε, λοιπόν, ε, τις εκθέσεις αξιολόγησης εξπόστε δεν τις παίρνει ούτε καν το Συμβούλιο, σαν και εμάς ενημερώνονται. Λοιπόν, προτιμώ αύριο στους συντονιστές να το συζητήσουμε το θέμα και όταν βρεθεί η λύση το συζητάμε. Εγώ είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένη από την επιστολή της κυρίας Δαμανάκη αλλά ε, και θεωρώ ότι δεν τηρείται η διαθεσμική συμφωνία. Λοιπόν, θα το παλέψουμε, θα συζητήσουμε αύριο όμως το θέμα. Για τις κομόρες τώρα. Εγώ βλέπω ότι αυξήθηκε κατά 27 ε, ε συγγνώμη παραγαδιάρικα, ε, ο αριθμός των σκαφών που είχαμε στη συμφωνία. Αλλά από την άλλη μεριά λέμε ότι ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν. Είχαμε μηδέν αλλιευτική δραστηριότητα. Λοιπόν, γιατί αυξάνεται ο αριθμός των παραγαδιάρικων. Λοιπόν, ε, υπάρχει κάποιο αίτημα του κλάδου, ο οποίος προηγουμένως δεν χρησιμοποιούσε τα παραγάδια και αποφάσισε να τα χρησιμοποιήσει τώρα. Ο κύριος Αλεξάνδρου έχει το λόγο. <clears throat> Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το γεγονός ότι μας παρουσίασε μια ολοκληρωμένη, ένα ολοκληρωμένο πίνακα ε, για το πρωτόκολλο αυτό. Εγώ ίδιος ε, έκανα την ε, διαπραγμάτευση και και πριν απαντήσω στις ερωτήσεις κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ε, ποιοτικέ σχέσεις που αυτό το πρώτο πρωτόκολλο ανεξάρτητα από την αλλιευτική ε, διάσταση και την ε, χρηματοοικονομική διάσταση λοιπόν την ποιοτική ε, διάσταση που έχει αυτό το πρωτόκολλο σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση που ακολουθούμε σε τέτοιες διαπραγματεύσει. Στο πρωτόκολλο αυτό περιλάβαμε μια ρήτα, ρήτρα αποκλειστικότητας, πάρα πολύ σημαντική, για να ε, περιλάβουμε τις δραστηριότητες όλων των σκαφών όταν ε, θέλουν να αλλιεύσουν στο αρχιπέλογο των Κομορών. Δεύτερη καινοτομία. Εισαγάγαμε μια ρήτρα αναθεώρησης που θα μας επιτρέψει να επανεξετάσουμε και να τροποποιήσουμε το πρωτόκολλο αν ε, απαιτηθούν ουσιαστικές ε, μεταβολές όσον αφορά τη στρατηγική της αλίας από πλευράς των ε, κομορών. Τούτο λοιπόν εμπίπτει στη στρατηγική της αλίας έτσι όπως ακολουθείται από τρίτες χώρες. Τρίτη καινοτομία και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντική που χρειάστηκε να διαπραγματευτούμε είναι ότι σαγάγαμε μια ρήτρα που επιτρέπει την διακοπή του πρωτοκόλου σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι το άρθρο 96 και του ε, άρθρου 9 της συνθήκης του Κοτονού. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια νέα διάσταση η οποία ε, εισάγεται και είναι διαφορετική από τα άλλα πρωτόκολλα τα οποία είχαν υπογραφεί στο παρελθόν. Και υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα διακοπής της ε, εφαρμογής του πρωτοκόλου ως προς την χρηματοδότηση εάν η πολιτική που ακολουθείται δεν εκπληρεί τους στόχους της. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, ε, κυρία Πρόεδρε, ότι αυτή ήταν μία από τις βαθιστικές αδυναμίες ε, των συμφωνιών που είχαμε συνάψει στο παρελθόν. Εκείνη την εποχή δεν είχαμε στη διάθεσή μας ρήτρε οι οποίες μας επέτρεπαν να διακόψουμε την ε, επαφή αν οι στόχοι δεν οι προϋποθέσεις δεν τηρούνταν. Τώρα λοιπόν με βάση τις νέες ρήτρες έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε από πιο κοντά τα πράγματα και να δούμε ότι αυτή η στήριξη κατά τομέα επιτυχάνει τους στόχους της. Τώρα, για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα στις ερωτήσεις ως προς την αύξηση του αριθμού των σκαφών. Υπάρχει πράγματι μια αύξηση ως προς τον αριθμό που εμφανιζόταν στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Αύξηση λοιπόν του αριθμού διότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις αλλιεύουσες χώρες. Παραδείγματος χάρη στο προηγούμενο πρωτόκολλο είχαμε 17 ε, σκάφη ενώ τώρα έχουμε 25. Είχαμε στο προηγούμενο πρωτόκολλο 25 ε, ήχο υποστηρικτικά. Και τώρα έχουμε ε, ε, και τώρα έχουμε 45. Από την άλλη έχουμε μία μείωση του, τον, του τονάζου αναφοράς, δηλαδή από 6.000 τόνους σε 4.850. Τούτο σημαίνει ότι αν Όλα αυτά τα σκάφη, όλα αυτά τα σκάφη ε, θα έπρεπε να αλλιεύουν, η μέση ποσότητα θα ήταν κατώτερη από τη μέση ποσότητα, αλλά αυτό σε θεωρητικό επίπεδο, ε, που θα εξασφάλιζαν σύμφωνα με το προηγούμενο πρωτόκολλο. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην ανησυχία που διατυπώθηκε από την κυρία Λαβίνα σχετικά με τα ηχθίδια. Και εμείς είμαστε ευαίσθητοι στο θέμα αυτό. Τη μείωση λοιπόν του τονάζου αναφοράς είναι ένα ε, βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας κυρία Πρόεδρε και αν υπάρχουν και άλλες είμαι έτοιμος να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. No, pero eso ya lo vamos a discutir mañana, así es que yo no quiero comentarlo con la comisión ahora. A ver, eh, señor Capoulas. Ο κύριος Καπώνης έχει το Νομίζω ότι αυτά που ακούσαμε μόλις από την Κομισιόν δεν απάντησαν στην ερώτηση που έθεσε η Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι αντικειμενικά απαντήθηκε η ερώτηση και ερμηνεύω το θέμα αυτού του ελάχιστου της ελάχιστης ποσότητας των παραγαδιών ως κομμάτι της προηγούμενης ε, ε, συμφωνίας να είναι ας πούμε αποτέλεσμα της πειρατείας ε, και να αλλάξουν τα πράγματα όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Επίσης, να σας ευχαριστήσω κυρία συνάδελφε που θέσατε το ζήτημα λεπτομερώς γιατί η σύνοψη που λάβαμε δεν δείχνει πόσο αναποτελεσματική είναι η... πόσο αναποτελεσματικός είναι ο έλεγχος και οι νέες ρήτρες στην επόμενη συμφωνία θα διασφαλίσουν ότι θα ε, βελτιωθούν αυτά τα προβλήματα και θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι ρήτρε, ειδικότερα όσον αφορά τον κλάδο της αλληλείας στις Κομόρες. Ειδικότερα όταν έχουμε υψηλότερο εισόδημα ανά άτομο, ειδικότερα για τους αλληλείς. Θέλουμε να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού και θεωρούμε ότι οι νέε ρήτρε θα βοηθήσουν και η αξιολόγηση θα είναι πιο θετική όταν αξιολογήσουμε πλέον αυτή τη συμφωνία και στη συνέχεια θα έχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες από την Κομισιόν, ελπίζω. Να πω στην πρόεδρό μας ότι υποστηρίζω πλήρως την πολύ σκληρή στάση που θέλει να τηρήσει αύριο στη συνάντηση των συντονιστών και στις συναντήσεις με την Επίτροπο γιατί η τρέχουσα κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δίκιο έχετε, αλλά σιγά σιγά πρέπει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, αυτή η ζώνη ελέγχεται από την CTO και εμείς ε, θα συμμετέχουμε στην ε, προπαρασκευαστική συνεδρίαση και θα γίνει πρόταση για ένα σύστημα ποσοστώσεων και η, Κομισιά, η Κομισιόν προσπαθεί να ενισχύσει σε αυτήν την ε, CTO τα διαχειριστικά μέτρα. Σε μερικούς μήνες θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, η συνάντηση. Ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο στην ημερήσια Α, συγγνώμη, ξέχασα την προθεσμία. 4 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και θα ψηφίσουμε τον Μάρτιο και θα πάει στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη και τώρα εγώ θα σας μιλήσω για την συμμετοχή μου ως παρατηρήτρια στην Χονολουλού τον Δεκέμβριο. Πήγα ως παρατηρήτρια στην συνεδρίαση και έρχομαι πραγματικά, επιστρέφω πάρα πολύ εντυπωσιασμένη από αυτήν την ε, συνεδρίαση. Και υπάρχει και μία έκθεση πολύ καλή της ε, Κομισιόν στη διάθεσή σας όπου αναλύονται όλα τα σημεία. Και εγώ όμως θα σας πω την προσωπική μου γνώμη για όλα αυτά. Λοιπόν, θα μακρηγορήσω, οπότε όποιον δεν τον ενδιαφέρει το θέμα να σηκωθεί να φύγει και να μείνει όποιος ε, τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, εγώ προτιμώ να μ' να μ ακούν αυτοί που ενδιαφέρονται και όποιον δεν τον ενδιαφέρει τίποτα να σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, έρχομαι εδώ πέρα. Με ένα πρόχειρο που το έχω εδώ μπροστά μου γιατί ήταν πριν από τις διακοπές. Εγώ που ασκώ κριτική πολύ συχνά στην Κομισιόν, όταν η Κομισιόν κάνει καλή δουλειά θέλω να τη το αναγνωρίζω. Ευχαριστώ λοιπόν την Κομισιόν για τη βοήθεια που μου δώσε για να μπορέσω να πάω. Το Συμβούλιο είχε πει ότι εγώ δεν μπορούσα να πάω διότι δεν είχα εκπληρώσει δεν ξέρω τι περίεργες προθεσμίες που έπρεπε να κρατήσω ενώ η Κομισιόν μου διευκόλυνε το ταξίδι. Τώρα κατά δεύτερο η Κομισιόν ήταν πραγματικά τέλεια. οι αρχηγοί της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερασπίστηκαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν έχουμε πολλά εκεί, έχουμε δηλαδή τέσσερα παραγαδιάρικα και ε, άλλα τρία λευτικιά, αλλιευτικά. Ε, Αλλά υπερασπίστηκαν τις αρχές ε, της υπεύθυνη και αηφόρου αλίας και ήταν δύσκολο για τον αρχηγό της αντιπροσωπείας να αντιπαρατεθεί έναντι χωρών οι οποίες ούτε καν θέλουν να ακούσουν τι θα πει η φορεία στην αλία, η υπεύθυνη αλία κλπ. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. 6 λοιπόν με 10 Δεκεμβρίου στην Χονολουλού η συνεδρίαση. Πρόκειται για την πιο πλούσια περιοχή του Ειρηνικού. Τα αλλιεύματα εκεί είναι το, είναι αντιπροσωπεύουν το 81% των αλλιευωμένων ειδών στον ειρηνικό και το 16% σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για παραμέτρους ε, που μη συγκρίσιμες. Το 9% είναι παραγάδια και όλο το υπόλοιπο είναι κανονική αλληλεία. 2.468.000 τόνοι ψάρια αλλιεύτηκαν στην περιοχή σύμφωνα με τα στοιχεία της περιοχής και αναφέρει τα αλλιεύματα η Πρόεδρος. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό σε αυτήν την συμφωνία είναι ότι εντάσσεται το 80% μέσα σε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, το άλλο 20% είναι νησιά. Ε, Παπούα, Μάρσαλ κλπ. που είναι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Αυτή είναι η ιδιομορφία αυτής της οργάνωσης και η σύμβαση φυσικά εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή, σε όλη τη ζώνη. Και να υπογραμμίσω για να συνειδητοποιήσετε πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση εκεί είναι ότι αυξήθηκε από το 2000 μέχρι σήμερα το, η αλλιεύσιμη ποσότητα και αυτό στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. <coughs> Μόνο η αλλιευτική προσπάθεια του στόλου αυξήθηκε σε τρία χρόνια από το 2008 μέχρι το 2011 κατά 40%. Δηλαδή η αύξηση της παράκτειας αλίας ήταν 40%. Και η κατάσταση των αλλιευτικών αποθυμάτων είναι ανησυχητική. Το, ε, τα αποθέματα του Skipjack μειώνονται πολύ σημαντικά. Είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση λοιπόν. Πόσο μάλλον ε, όταν ε, ε, βρίσκονται υπό ναυπήγηση άλλα 40 πλοία. Δηλαδή προχωράνε πράγματα αντί να περιορίζονται. Ενώ έχει ζητηθεί μείωση της αλλιευτικής προσπάθειας κατά 39% και βλέπουμε όμως αντίθετα ότι έχουμε αύξηση 40%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κράτη που απαρτίζουν τη συμφωνία είναι μικρά νησιωτικά κράτη και θα το επιβεβαιώσει αυτό και η Κομισιόν και δεν θέλουν την αηφόρο αλία με δύο προσχήματα αφενός ένα το αναπτυξιακό στοιχείο αυτό βαντεσουά που λένε οι Γάλλοι είναι αυτονόητο και δεύτερο που είναι πολύ πιο σοβαρό είναι ότι θεωρούν ότι οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται στην πόδα αυτή θα πρέπει να αφορά μόνο την περί τα διεθνή ύδατα. Έχουμε την creeping jurisdiction στα αγγλικά όπου θεωρούν ότι στις ε, ζώνες, ε, στις ε, ΖΕΕ δεν, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η σύμφωνία αυτό που αποφασίζει η πόδα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε εκεί πέρα. Διότι κάθε φορά. Που πάει να περάσει ένα μέτρο λένε όχι, όχι, στα χάησης εφαρμόζεται, δηλαδή στην ανοιχτή θάλασσα εφαρμόζεται, στα διεθνή ύδατα, όχι σε εμά. Και οι θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη Ιαπωνία. δεν εισακούγονταν γιατί είναι οι μικρές νησιωτικές περιοχές. Αλλά εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα βλέποντας τη στάση της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας και επειδή έχω καλή ανατροφή δεν θέλω να χαρακτηρίσω τη συμπεριφορά τους αλλά έμεινα άναυδη. Και δεν καταλαβαίνω η Νέα Ζηλανδία η οποία πάει σε όλα τα φόρα και φωνάζει περί αηφορία στην Αλία εκεί πραγματικά το βούλωσε και κράτησε ένα χαμηλό προφίλ ενδίδοντας στις θέσεις αυτών των μικρών χωρών. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θέλουν να είναι σύμμαχοι αυτών των μικρών χωρών. Κατά δεύτερο, να σας πω ποια είναι τα πιο συγκεκριμένα αυτής της συνεδρίασης. Και τι μας οδήγησε δηλαδή σε μια τέτοια παράδεκτη κατάσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στα στοιχεία. Κανένας εκεί δεν στέλνει στοιχεία ή οποιαδήποτε έκθεση. Δύσκολα λοιπόν κανείς μπορεί να διασφαλιστεί ότι εκεί τα ελάχιστα μέτρα τα οποία ισχύουν τηρούνται. Πάμε στο επόμενο σημείο. Τα... Στα Port State Measures πρόκειται για ένα μέτρο που έχει τη ρίζα του στην ΦΑΟ, στην... Και κάθε φορά που μιλάνε για αυτό το πρόβλημα, σε αυτή την περιοχή του Ινδικού αναφέρονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είχε μία πρόταση η οποία ήθελε να θέσει σε λειτουργία όλα αυτά τα μέτρα τα σχετικά με τα λιμάνια για να καταπολεμήσει την πλά. Την αλία είναι. Υπήρξε μία πλήρης αντίρρηση. Κανένας δεν ήθελε αυτά τα εφαρμοστικά μέτρα και είπαν ότι δεν θα τα εφαρμόσουν ούτε καν στα, εξω... στα αλλοδαπά σκάφη τα οποία ψαρεύουν στην περιοχή ούτε στα δικά του σκάφη φυσικά δηλαδή στις ε, ΑΟΖΑ δεν δέχονται την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε μία πρόταση για το Catch Documentation Scheme, δηλαδή τα βασικά και ουσιαστικά στοιχεία για την καταπολέμηση της ε, αλίας της παράνομης αλίας. Και είχαμε την υποστήριξη για την ΠΛΑ ε, και για τη Ιαπωνία κλπ. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι άμα δεν τηρηθούν οι όροι της Catch Documentation Skin για την πλά, αυτές οι χώρες στο μέλλον δεν θα μπορέσουν να εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ο κανονισμός ε, για την αλλή απλά 2005-2006 εγγυάται ότι τα αλληλεύματα που έρχονται στην Ευρώπη δεν θα, είναι, δεν θα πρέπει να είναι αλλιεύματα πλά. Και εγώ το αναγνωρίζω ότι είμαι κακιά κάκιστη. Η παππού Νέα Γουινέα ήταν αυτή η οποία έφερε και τις μεγαλύτερες αντιρρήσεις. Η παππού Νέα Γουινέα η οποία προεδρεύει του FFA είναι ένα από τα φόρα που έχουν εκεί είναι μία από τις χώρες η οποία αρνήθηκε την εφαρμογή της Catch Documentation Scheme. Γι' αυτό σα το λέω επειδή είμαι κακιά πολύ κακιά. Και το γεγονό ότι η παππού Ανέγου, η Νέα δηλαδή δηλαδή 20 κεφάλι μετά από όλε τι συζητήσεις που είχαμε εδώ ε, πραγματικά με τσάτισε. Και να σας πω και το άλλο δηλαδή που δεν πίστευα τι άκουγα στα αυτιά μου. Υπήρχαν ένα πρόγραμμα το οποίο ελέγχεται από τα συμβαλόμενα μέρη και όχι συνολικά. Και ζήτησε η Ιαπωνία να σταλούν οι εκθέσεις των παρατηρητών. Και η Κομισιόν και η Ιαπωνία είπανε ότι όταν σε κάποιο από τα προβλήματα εμπλέκεται ένα κοινοτικό σκάφος πρέπει να ξέρουμε τι συνέβη για να μπορέσουμε να εργαζόμαστε εκεί. Προς μεγάλη έκπληξη των πάντων αυτές οι χώρες μεταξύ των οποίων και η Παππούα Νέα Γουινέα είπανε ότι αυτό το θέμα και, και να σας τα πω αγγλικά δηλαδή είπαν ότι είναι domestic business διότι εκεί μόνο αγγλικά μιλάνε και δεν αφορούσαν σε κανέναν από τα συμβαλλόμενα μέρη. Και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επανήλθε και επέμεινε στη γραμματεία της Διεθνούς Επιτροπής Αλίας είπε ότι εγώ δεν έχω πάρει ποτέ καμία έκθεση παρατηρητών. Φαντάζεστε τι έγινε. Και είπανε ότι στα δικά τους χωρικά ύδατα δεν έχουν να στέλνουν καμία έκθεση. Και μείναν όλοι άναυδοι. Όχι μόνο δηλαδή δεν δίνουν την έκθεση στα συμβαλόμενα μέρη, αλλά το δίνουν ούτε στην Western. Πραγματικά εγώ δεν το καταλάβαινα πια αυτό το χάος και μίλησα με έναν ε, Ισπανό εφοπλιστή που είχε ένα σκάφος εκεί και είπαν καλά ε, παιδιά εσείς πώς λέγετε και μου είπε κοίτα να δεις Κάρμεν εγώ πρέπει να στέλνω έναν παρατηρητή για τα χάισις, για την ανοιχτή θάλασσα, για το πέλαγος και άλλο παρατηρητή όταν μπαίνω στην πόδα τι μία χώρα εκεί. Κανένας λοιπόν δεν είναι ενήμερος για το τι συμβαίνει. Και πάω τώρα στο δεύτερο, για τον έλεγχο χωρητικότητας των α, λιευτικών. Οι Ιάπωνες ήρθαν να με βρούνε για να ζητήσουν ευρωπαϊκό έλεγχο για τα λιευτικά στην περιοχή. Και η Ιαπωνία παρουσίασε μία πρόταση λέγοντας ότι σε την πόδα δεν γίνεται τίποτα από τα συμφωνημένα ότι αυξάνεται η αλληλευτική ικανότητα αντί να παγώνει δεν πληρούμε εμεί τους στόχους ε, της ε, πόδα και θα έπρεπε να θέσουμε να κάνουμε εμεί μία πρόταση που να σταματάει το θέμα της χωρητικότητας. Και είπε βέβαια η Ιαπωνία επειδή έχουμε εδώ πέρα πολλές αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει σίγουρα να βρούμε μία μεγαλύτερη ευελιξία για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υποστηρίχθηκε η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τον Καναδά αλλά αυτές οι χώρες της πόδα μεταξύ των οποίων και Παππούα Νέα Γουινέα είπαν καθαρά και εξάστερα ότι η μείωση της αλληλευτικής τους ικανότητας δεν ήταν λύση και είπανε ότι αυτό θα γινόταν σε βάρος των αναπτυσσομένων χωρών. Συγίνει χθίως η Αυστραλία. Και η Παππούα Νέα Γουινέα που κατέκρινε περισσότερο από όλους την πρόταση και η Ιαπωνία είπε στην Παππούα. Τους είπαν κοιτάστε εσείς έχετε καμιά τρενταριά δικά σας σκάφη. Αλλά έχετε όμως και πολλούς προσκεκλημένους ε, στη δική σας ε, πόδα. Και όσοι ασχοληθήκατε με την Παππούα Νέα Γουινέα ξέρετε πολύ καλά σε τι αναφέρομαι. Τους είπε η Ιαπωνία You have too ε, many guests in our waters. Έχετε πολλούς ε, προσκεκλημένους ε, στα ύδατά σας. Αλλά αντί όμως να περιορίσουν τις ελληνικές ικανότητες και μετά και τα νησιά Μάρσαλ, ψάξτε τα στο χάρτη γιατί έτσι με πρώτη ματιά δεν τα βλέπετε, είπανε ότι θα ναυπηγήσουν τέσσερα νέα σκάφη και κάθε αλλιευτικό σκάφος ισχύει 20 ε, κοστίζει 20 εκατομμύρια δολάρια. Θα μου πείτε ποιος τα πληρώνει όλα αυτά. Γιατί τα νησιά Μάρσαλ δεν έχουν λεφτά να τα πληρώσουν. Εγώ ξέρω ποιος τους τα πληρώνει βέβαια. Και εσείς το ίδιο. Η να ναυπηγεί αλλιευτικά σκάφη ασταμάτητα και όταν δεν έχει πια άλλα περιθώρια για δική της νεολόγηση, δική της σημαία, τότε τα να πηγεί με τη σημαία αλωνών. Και αυτή η συζήτηση λοιπόν έμεινε άκαρπη και συνεχίζουν να μην λαμβάνουν να λαμβάνουν κανένα μέτρο και να ολοκληρώνω πριν από τα τελικά πολιτικά μου συμπεράσματα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε μία πρόταση για την μείωση της προσπάθειας σε όλη τη ζώνη, αλλά αυτό μόνο για τα χάησης. Ζήτησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλειστεί η περιοχή για τρεις μήνες και βεβαίως οι χώρες, οι μικρές χώρες είπανε κουβέντα να μην γίνεται. Εγώ ήρθα πραγματικά ιδιαίτερα ενοχλημένη από όλη αυτή την συνεδρίαση. Πρόκειται λοιπόν για μία μειοψηφία η οποία δεν καταφέρνει πραγματικά τίποτα. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς ε, να σμπρώξουμε αυτές ε, τις χώρες να κάνουν κάτι Και πρέπει να μας πει η Επίτροπος τι θα κάνει με όλες αυτές τις χώρες και με τα πιστοποιητικά αλίας αυτών των χωρών. Δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι ό,τι έρχεται από εκεί δεν είναι πλά. Διαβάζω εγώ και πάλι τον κανονισμό 1005 ε, όπου λέγεται ότι οι πόδα, που δεν συμμετέχουν σε μία αηφόρα διαχείριση να τις αποφεύγουμε. Και το λέω όχι για να τους ζημιώσουμε, γιατί το καταλαβαίνω πολύ καλά ότι είναι αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά αυτές οι χώρες να συνειδητοποιήσουν ότι εκεί θα πρέπει να δρουν με άλλο τρόπο, διότι αυτή η περιοχή του Ειρηνικού που είναι η πιο πλούσια από όλους, θα καταστραφεί δεν είναι μόνο ο ρόλος μας να πάμε εκεί και να είμαστε και άψογοι στην παρουσία μας, αλλά να ληφθούν και μέτρα ώστε αυτές οι χώρες να πάρουν τα πράγματα στα σοβαρά, διότι δεν θα το λάβουν ποτέ υπόψη τους το θέμα. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και θα πρέπει να έχουμε και κάποια αντίπεινα ούτως ώστε καλού, με το καλό ή με το κακό να τους υποχρεώσουμε να λάβουν μέτρα για μια πιο εφοροαλία. Εγώ είδα μια τεράστια παθητικότητα πάντως Λοιπόν, παθητικότητα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν θέλουν να αντιπαρατεθούν σε χώρες οι οποίες λένε είμαστε φτωχές και είμαστε αναπτυσσόμενοι. Αλλά εντάξει, φτωχοί είναι τώρα άλλο να είσαι φτωχός και βλάκας και άλλο φτωχός και μόνο. Τώρα εμείς τέσσερα λιευτικά έχουμε εκεί και τέσσερα παραγαδιάρικα. Δεν έχουμε τίποτα το φοβερό, τέλος πάντων. Μακρηγόρησα και μπορεί να ήμουν και βαρετή. Αλλά πραγματικά ήθελα να σας εκφράσω το αίσθημά μου, γυρνώντας από εκεί, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό για να μην το πάρουμε στα σοβαρά και συνδέεται και με άλλες ε, πτυχές όπως αυτή η περίφημη συμφωνία που ψηφίσαμε τις προάλλες. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται και πολιτικά θα πρέπει να λάβουμε στο μέλλον αποφάσεις. Και τέλος πάντων όλα αυτά ήταν καθαρά και εξάστερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας έκανα αυτή την παρουσίαση. Η κυρία Αντρές Μπαρεά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που εξηγήσατε με πάθος το πώς ε, έγιναν οι συζητήσεις. Υπάρχουν θέματα που με ανησυχούν σχετικά με τα όσα μας είπατε και ειδικότερα για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μας είπατε ότι η Κομισιόν ήταν πολύ θετική σχετικά με αυτά που είδατε και παρατηρήσατε. Έκανε, έβγαλε μία έκθεση η οποία την οποία διάβασα και αξιολόγησα πολύ προσεκτικά. Μας είπατε επίσης ότι η Κομισιόν θέλει να προσπαθήσει να επιλύσει τα προβλήματα που περιγράψατε, τα οποία είναι σημαντικά και σοβαρά. Στην Ολομέλη της Προάλλες, πραγματικά υπόθηκε μια πολύ σωστή άποψη. Ακούσαμε από την Κομισιόν ότι δεν υπάρχει έγγραφο το οποίο να λέει ακριβώς αυτά που είπε η Κομισιόν στην Ολομέλεια της προάλλες. Ουσιαστικά όμως δεσμεύτηκε για μία έκθεση αξιολόγηση ε, για την κατάσταση στην περιοχή αυτή. Είπε βέβαια ότι όλα ήταν υπό έλεγχο, δεν υπήρχαν ε, προβλήματα και τα πράγματα εξελίσσονταν σωστά. Εδώ υπάρχει μάλλον μια αντίφαση και νομίζω ότι πρέπει να διαλευκάνουμε το θέμα. Να δούμε. Αν όλα αυτά που μόλις είπατε ισχύουν. Ε, πώς αυτό συμβιβάζεται με αυτά που είπε η Κομισιόν της προάλλες στην Ολομέλεια όταν η Κομισιόν μας λέει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στην περιοχή. Μάλλον μια... ένας διχασμός απόψεων υπάρχει εδώ μεταξύ της Κομισιόν και της υπόλοιπης Επιτροπής και μάλλον χρειάζονται διευκρινήσεις ίσως ε, να υπάρχει ε, έλλειψη συμφωνίας εντός της ίδιας της Επιτροπής. Κυρία Λέβεν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Φρέρ, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θα ήθελα κι εγώ να πάω στη Χονολιλού, αλλά πολύ αργά το σκέφτηκα μάλλον. Γνωρίζω όμως πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν ενεργό ρόλο στη διεθνή αρένα, ειδικότερα όχι μόνο για την πλά, αλλά, που ήταν η έκθεσή μου, αλλά και για την ε, πρόθεση της βιώσιμης αλληλείας ε, που σε συνδυασμό με την Ιαπωνία και τις Ηνωμένε Πολιτείες προσπαθούν να την προωθήσουν. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερο δυναμικό από ό,τι άλλες δύο υπερδυνάμεις στην αλληλεία γιατί εκείνες περισσότερα κοιτούν να είναι προστατευτικές παρά να έχουν μια πιο παγκόσμια θεώρηση των πραγμάτων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κανόνες ε, των ΠΟΔΑ. Και πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε, γιατί αν έχουμε συμφωνίες της ΠΟΔΑ οι οποίες δεν μεταφράζονται σε εθνική νομοθεσία δεσμευτική σε εθνικό επίπεδο, τότε είναι άχρηστες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα από τα κύρια σημεία που πρέπει να δούμε σε όλα τα σε όλες τις πόδα στον κόσμο, στην ICAT και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχουμε αυτό το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φανταστείτε πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση ε, γνωρίζω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Lace Act για την παράνομη αλληλεία ε, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Εάν το σκάφος έχει παραβιάσει έναν κανόνα της πόδα, αλλά όχι εθνική νομοθεσία, τότε δεν θεωρείται παράνομη αλληλεία. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα και υπάρχουν πολλές επιπλοκές θα έλεγα και γι' αυτό θα έπρεπε να είναι ύψης της προτεραιότητας ε, η προσπάθεια να πείσουμε τα κράτη να εφαρμόσουν τους κανόνες των ποδα... Η είναι άχρηστη. Η ιδέα των πολιτικών εισαγωγής-εξαγωγής που θέσατε κυρία Φράγκα είναι ενδιαφέρουσα. Ελπίζω να συνεισφέρετε στη συζήτηση για την έκθεσή μου ε, που αναφέρονται όλες αυτές οι ιδέες ε, γιατί χρειάζεται να έχουμε όλα τα έθνη σε αυτή τη συζήτηση για να έχουμε όχι μόνο ε, νόμιμη αλληλεία και βιώσιμη αλληλεία. Να πω ότι είπα σήμερα το πρωί για τους παγκόσμιους ωκεανούς που είναι η παγκόσμια κληρονομιά και για τη σπόδα. Ε, υπάρχουν ε, μικρά και μεγάλα έθνη που καταστρέφουν τους ωκεανούς και στον βαθμό που αναφέρατε με την ε, υπερβολική δυνατότητα ναυπήγησης νέων πλοίων 40% αύξηση ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μείωση 40% πώς οι μελλοντικέ γενναίες θα αποδεχτούν ότι τα βλέπουμε όλα αυτά και δεν κάνουμε τίποτα έχω συζητήσει πολύ και σκεφτεί σε συνεργασία με ανθρώπους που ασχολούνται με τη διεθνή νομοθεσία. Όμως θεωρώ πως αυτό το θέμα πρέπει να μπει στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης και να υπάρχουν ανεξάρτητες αξιολογήσεις των πόδα μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ ίσως. Ε, ίσως η δημιουργία νέου φορέα στον ΟΗΕ που θα αναλάβει την ευθύνη για την απόδοση των πόδα και την έκδοση ανεξάρτητων εκθέσεων έτσι ώστε να μπορεί ως επόμενο βήμα να υποχρεώσει τις χώρες των ΠΟΔΑ να αναλάβουν δράση και να εφαρμόσουν αυτά που συμφωνούνται, ίσως να είναι το ε, απαραίτητο. Και μετά πάμε στο επόμενο πρόβλημα της λήψης αποφάσεων στις ΠΟΔΑ. Είπαμε ότι στις περισσότερες υπάρχει ένα συνενετικός τρόπος λήψης αποφάσεων. Όταν κάποιος δεν φέρεται σωστά, θα πρέπει να συμφωνήσει να υποστεί κυρώσεις. Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε περισσότερο αύριο όταν παρουσιάσω το έγγραφο εργασίας για τη ΣΠΟΔΑ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρόλα αυτά. κύριος, κυρία Ρόδος. Ναι, ευχαριστώ και εγώ να σας ευχαριστήσω κυρία Φράγκα θερμά για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεσή σας. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα. Όχι μόνο αυτά ε, για τα οποία μας πληροφορήσατε, για το τι συμβαίνει στον κόσμο, όπως είπε και η κυρία Λέβεν, αλλά υπάρχει και το άλλο εσωτερικό πρόβλημα. Όταν μιλάμε για την πολιτική ανάπτυξη και με τον Επίτροπο που είναι υπεύθυνο συζητούμε, όταν συζητούμε έχουμε άλλη ενημέρωση. Τι γίνεται με τη κοινή στάση λοιπόν που πρέπει να έχουμε εδώ. Ίσως θα πρέπει να προσκαλέσουμε και τους δύο επιτρόπους γιατί σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν στην Ολομέλεια και από τον κύριο Μάρτιν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όμως ε, αυτά που μας είπατε είναι διαφορετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει εσωτερικά να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από κοινού. Και αυτό είναι αδυναμία όταν δεν πηγαίνουμε αποφασισμένοι στις διεθνείς μας δράσεις. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε με, τους, ε, με την Κομισιόν, τους πολιτικούς και τους βουλευτές που ασχολούνται με την πολιτική ανάπτυξη για να δούμε πώς ε, θα τηρούνται οι συμφωνίες, πώς θα γίνονται οι κυρώσεις και όλα αυτά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ευχαριστούμε για την πολύ ξεκάθαρη παρουσίαση. Και για το γεγονός ότι μας ενημερώσατε για μια κατάσταση η οποία είναι άκρος ανησυχητική. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Εσείς μιλήσατε για μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε ε, πιστοποιητικά εξαγωγών. Ερώτημα. Ποιο είναι το ποσοστό των εξαγωγών που δεχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που αλλιεύονται σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε δηλαδή χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες και με τις συμφωνίες μπορούν να συνεχίσουν να πράττουν ό,τι επιθυμούν ή μπορούμε ας πούμε να ακυρώσουμε τις, ε, τα πιστοποιητικά που έχουν ή τις άδειες που έχουν και να μην εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ναι, ε, εδώ υπάρχουν διάφορα θέματα. Πρώτον, πώς αυτές οι πόδα λειτουργούν και τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μπορεί να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ε, πρώτα απ' όλα μία μειοψηφία αυτών των χωρών έχουν ε, βιώσιμη αηφόρο αλία. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Ε, τις προάλλες, ο Επίτροπος Ανάπτυξης ο, μιλούσε περί του εμπορίου και ουσιαστικά πρόκειται για θέμα εμπορίου. Αυτό ελέγχθηκε άλλωστε και στη διάσκεψη. Ε, ο Επίτροπος είπε ότι οι εφοπλιστές, οι ιδιοκτήτες των σκαφών ή μάλλον να το πω αλλιώς, η ευρωπαϊκή πλευρά των πλειοκτητών δεν έχει θέσει κανένα ζήτημα. Και ο κύριος Δεμπρούχο, ο Επίτροπος, δεν μίλησε καν για τον τομέα αλίας της Ευρώπης, δεν Είπε λοιπόν ο Επίτροπος, η Κομισιόν επιδιώκει να απελευθερώσει την, τον τομέα των εξαγωγών αλίας και αυτό είναι όλο. Δηλαδή εδώ υπάρχει παντελή έλλειψη συντονισμού κάποιες χώρες, τρίτες χώρες έχουν δικαιώματα για την ανάπτυξη, ε, για την πρόθεση της ανάπτυξής τους, για την πρόθεση των εξαγωγών τους κλπ. Ωστόσο, εάν κοιτάξουμε τους κανόνες, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται τα πράγματα φαίνεται να οδηγούν ότι οι πάντες είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν από την Ιαπωνία μέχρι την Παππούα Γουινέ, που οδηγεί σε μία μη βιώσιμη αλία. Υπάρχει δηλαδή ένας πλήρης, μια μη βιωσιμη αλληλεια έλλειψη συντονισμού μεταξύ των στόχων της ανάπτυξης και του στόχου της απελευθέρωσης. Δεν υπάρχει συντονισμός και πρέπει να γίνει κάτι, τουλάχιστον στο επίπεδο της αλληλείας και αυτό δεν γίνεται. Διότι ο καθένας δουλεύει στο δικό του τομέα και αφενός έχουμε την Κομισιόν που λέει απελευθέρωση των εξαγωγών για τις χώρες αυτές και βεβαίως τούτο αφορά και στα ε, ψάρια και από την άλλη λέμε ε, βιώσιμη η αηφόρο αλία. Αυτά τα δύο δεν είναι συμβατά. Αν κοιτάξουμε τώρα τα επεξεργασμένα ε, προϊόντα, μεταποιημένα προϊόντα, η Παππούα Νέα Γουινέα είναι μεταξύ των έξι χωρών που εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, είναι σαφές και το ακούσαμε και στην Ολομέλεια της προάλλες, είναι σαφές ότι όσον αφορά την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της συμφωνίας με την Παπούα, Νέα Ουινέα και τα Φίτζι, θα πρέπει να υπάρξει άρδιν αναθεώρηση των κανόνων προέλευσης που ισχύουν. Έχουμε εκθέσεις από την Γενική Διεύθυνση 12, αλλά νομίζω ότι δεν έχει γίνει μια μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων ε, στο γενικότερο τομέα της αλληλείας στην περιοχή και μπορούν οι χώρες αυτές να εξάγουν ελεύθερα χωρίς κανέναν περιορισμό. Όταν λοιπόν συζητούμε τι είδους μελέτες θέλουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε μία μελέτη στόχων για να μας δώσει μία σφαιρική εικόνα της κατάστασης περιλαμβανομένων των πληροφοριών από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και από την ε, Διεύθυνση Αλίας. Δεν είχαμε μέχρι τώρα σωστή ανάλυση επιπτώσεων που να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές, όλες τις επιπτώσεις. Έλλειψη λοιπόν συντονισμού στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμπλέκονται οι διάφοροι επίτροποι, εμπλέκονται διευθύνσεις, αλλά δεν υπάρχει συντονισμός. Ο κύριος Ντεγκούχτη ήθελε να ασχοληθεί με το θέμα της προάλλης, με μια άλλη ευκαιρία και είπε ότι υπάρχουν προβλήματα στην Αλία, αλλά δεν ήταν σε θέση να αναφερθεί λεπτομερώς στα προβλήματα αυτά. Θα το Αυτό επιβεβαιώθηκε στην συζήτηση. Το 90% των παρισταμένων ήταν μέλη που είχαν άμεσο συμφέρον στην Αλία. Αλλά ο κύριος Ντεγκούχτ δεν ήθελε να απαντήσει σε ερωτήσεις σε κανένα θέμα, γιατί πίστευε ότι πάνω από όλο αυτό που είναι σημαντικό είναι η απελευθέρωση των εξαγωγών των αλληλευτικών προϊόντων. Αυτό είναι όλο. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι παγκοσμίως τα παγκοσμίω το θέμα της αλίας βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά ε, στην ατζέντα και το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη είναι, υπάρχουν οι Ιάπωνες και άλλοι ε, ισχυροί ενδιαφερόμενοι από τον ειρηνικό που μπαίνουν στο παιχνίδι. Το, τα, τα βάρη, τα τονάζ είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Και όταν η Παππούα Νέα Γουινέα αντιτίθεται με το πάγωμα της, ε, ε, του όγκου ε, της παραγωγής της, αυτό γίνεται απολύτως αντιληπτό. Ο καθένας θέλει να κάνει την μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της ΑΟΣ του. Αλλά ο ειρηνικός είναι μια πολύ πλούσια περιοχή. Αλλά άμα συνεχίσουμε με τέτοιου ρυθμού, σε δύο-τρία χρόνια η κατάσταση θα γίνει καταστροφική. Ε, έχουμε ακόμη καιρό για να αντιδράσουμε. Εμείς λοιπόν πολιτικά έχουμε επιχειρήματα να το προβάλλουμε το θέμα στον, στην Επίτροπο αλλά πραγματικά είναι ανησυχητικό ο κύριος Ντεγκού επιτρέπει μέσα από παρεκκλήσεις Ε, χωρίς ε, ε, με, δασμό μηδέν τέλος πάντων και η... τελείωσα και τελειώνουμε μέχρι τις τρεις ακρόαση για την Ισλανδία και να είστε παρόντες πέρα στη συνεδρίαση